υπάρχει και απειλή στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της χώρας. Χαιρετίζουμε την ειρηνευτική συμφωνία που υπογράφηκε στις 11 Ιανουαρίου στο Λιμπρεβίλ και καλούμε τα μέρη να τηρήσουν την, ε, ε, την κατάπαυση του πυρός λαμβάνοντας υπόψη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί βλέπουμε ότι στρατολογούνται όλο και περισσότερα παιδιά στρατιώτες και υπογραμμίζουμε την ανάγκη για ασθενή παρακολούθηση της περιφερειακής διάστασης της σύγκρουσης. Επίσης τώρα θα στείλουμε μια αντιπροσωπεία ντρουά στην Αιθιοπία και θα κάνουμε και μια ανταλλαγή απόψεων για μια ολόκληρη μέρα με την Αφρικανική Ένωση. Πολλά από αυτά τα ψηφίσματα λοιπόν και οι καταστάσεις συγκρούσεων στην Αφρική θα συμπεριληφθούν στον κατάλογο των συζητήσεων που θα έχουμε στην Αντίσα ε, εγκρίναμε επίσης ψήφισμα κατεπήγοντος για την Ινδία τον Ιανουάριο ε, και επίσης ε, έχουμε και κατά του Ντάλιτς το Δεκέμβριο έχουμε εγκρίνει ένα ψήφισμα. Έχουμε λοιπόν δύο διαδοχικά ψηφίσματα που αφορούν την ανάγκη η κυβέρνηση της Ινδίας να αντιδράσει, να αντιδράσει πιο έντονα. πρέπει να δούμε πώς παρακολουθούν αυτά τα κατεπήγοντα θέματα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Αυτό έχει, αφορά όλα τα κατεπήγοντα. Και στο Κοινοβούλιο νομίζω ότι πρέπει να δούμε πώς θα βελτιώσουμε και θα παρακολουθούμε καλύτερα και αποτελεσματικότερα τα κατεπήγοντα αυτά θέματα. Επίσης εγκρίναμε ψήφισμα για την κατάσταση στο Μπαχρέιν αλλά νομίζω ότι θα επανέλθουμε σε αυτό όταν ακούσουμε τη σχετική έκθεση από την αντιπροσωπεία που πήγε στο Μπαχρέιν. Αυτό δεν ήταν όμως επίγον. ήταν ένα στεναρό ψήφισμα του Κοινοβουλίου σχετικά με τους πολλούς θανάτους ε, εργαζομένων στα κλωστοϊφαντουργία του Μπαγκλαντές. Και ζητούμε από την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές και στο ψήφισμα αυτό, όπως και ζητούμε από την κυβέρνηση του Πακιστάν, να κάνει ενδελεχείς έρευνες σχετικά με τις, τα πρόσφατα γεγονότα και να ε, λάβει μέτρα για να προλάβει την ε, επανάληψη αυτών των ε, θανάτων. Επίσης, αναφέρουμε την ευθύνη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που λειτουργούν στο εξωτερικό και ζητούμε από τις αρχές του Μπαγκλαντές να ερευνήσουν ειδικότερα το βασανισμό και δολοφονία του Αμίν Αλ ακτιβιστή για τα δικαιώματα εργασίας και να άρουν τους περιορισμούς στη συνδικαλιστική δράση και στις συλλογικές διαπραγματεύσεις στη χώρα αυτή. Ο συνάδελφος Λάιχτριντ από την ομάδα των Σοσιαλιστών Δημοκρατών παρουσίασε τεκμηρίωση από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ιανουαρίου 2013 σχετικά με το, τον ακτιβητή Σιράμι Μπανταρανεγιάκη, ο οποίος είναι ε, ανώτερος δικαστής στη Σρι Λάνκα, ο οποίος απομακρύνθηκε από το αξίωμά του. Ε, θα πρέπει να παρουσιάσει το, την αιτιολόγηση. Ε, τώρα υπάρχει όμως και ε, διαδικασία απόδοσης ε, κατηγοριών στον ε, δικαστή από το μεγαλύτερο κόμμα της χώρας. Εγώ εξέφρασα ανησυχίε ότι αυτή η διαδικασία απόδοσης κατηγοριών προσαγωγής έχει πολιτικά κίνητρα και επίσης Αναφέρομαι και στον Άβε Πιλαή που είναι είπατη εκπρόσωπος ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα ο οποίος ε, αναφέρει ότι πρόκειται για μεγάλη οπισθοδρόμηση στο κράτος δικαίου. Σήμερα στη Σρι Λάνκα η, Ένωση, η μεγαλύτερη Ένωση Δικηγόρων είπαν ότι θα μποϊκοτάρουν τον ε, καινούριο επικεφαλής του δικαστικού σώματος. Αυτά έχω να σας πω για την υπόθεση. Θα ακούσουμε περισσότερα για τη Σρι Λάνκα όταν πάμε στην Γενέβη, στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ε, στη Σρι Λάνκα ε, υπήρξε και μια ε, ε, στη Σαουδική Αραβία μια υπήκοση στη Σρι που αποκεφαλίστηκε δούλευε εκεί και ήταν στη φυλακή από το 2007 η Κάθριν Άστον νομίζω και ε, ε, εμείς διαμαρτυρηθήκαμε ε, για την εκτέλεση αυτή και τη θανατική ποινή γενικότερα και ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Σαουδικής Αραβίας ταξιδεύει στην Ευρώπη και ζήτησε να μας δει. Οπότε αξιοποίησα την ευκαιρία, η συνάντηση ελπίζω να γίνει και θα μιλήσουμε και για άλλα θέματα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σαουδική Αραβία. Μια άλλη καταδίκη θανατική έλαβε χώρα στο Μπαγκλαντές ε, για έγκλημα πολέμου. Ε, το Διεθνές Πυρηνικό Δικαστήριο στην Μπαγκλαντές ε, ε εκδίκασε την υπόθεση από το 1971. Ήταν μια καλή δίκη για να συζητηθεί και για να καταλήξουν και σε αποφάσεις, όχι όμως να επιβάλλουν τη θανατική ποινή. Και πάλι η Λέδη Άστον διαμαρτυρήθηκε κατά της εκτέλεσης αυτής. Η Βαρόνη Άστον επίσης έκανε δημόσια δήλωση και καταδίκασε την εκτέλεση έξι ανθρώπων στην Ταϊβάν. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα αύριο στην ώρα των ερωτήσεων. Τέλος, ε, είχα μία συνάντηση με την ε, Νάβε Πιλάη, ε, υπεύθυνη για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ήταν στις Βρυξέλλες και με διαβεβαίωσε ότι επίσης παρακολουθεί το έργο των θεσμικών οργάνων της Ένωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Επιτροπή μας. Χαίρεται διότι ε, είπα τι εκπρόσωπος στις Βρυξέλλες ε, την ενημερώνει συχνά. Ε, για την Ευρώπη λέει συχνά ότι το πώς αντιμετωπίζουμε τους Ρώμα το δικαίωμα των ετούντων άσυλο, αλλά και συγκεκριμένες καταστάσεις χωρών όπως ε, ε Σουδάν κλπ. Ε, μελετώνται από τους υπεύθυνους. Θα με στην Γενέβη, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αντιπροσωπεία και ελπίζω την, να συναντήσω πάλι την ε, κυρία Πιλάη. Επίσης υπογραμμίζουμε πόσο σημαντι Είναι σημαντική η δουλειά μας, μας είπε, γιατί αντικατοπτρίζεται και στα αποτελέσματα από τις μελέτες των Ηνωμένων Εθνών. Υπάρχουν περιοδικές ανασκοπήσεις της κατάστασης στη Γενέβη και μετά εξετάζουμε τις συστάσεις και κάνουμε και συνεδριάσεις εδώ. Γιατί έτσι ε, ε, έχουμε και αριστής ποιότητας ενημέρωση. Ευχαριστώ λοιπόν που με ακούσατε και τώρα Περνάμε στο επόμενό μας θέμα. Θα μας ε, ενημερώσει η αντιπροσωπεία Ντρουά που πήγε στο Μπαχρέιν από 18 μέχρι 21 Δεκεμβρίου. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλό ότι είχαμε στενή συνεργασία με την πρεσβεία στο Μπαχρέιν για να προετοιμάσουμε την επίσκεψη και έτσι η αντιπροσωπεία ε, μπόρεσε να κάνει πολλές συναντήσεις να δει την κατάσταση επιτόπου που σε κάποια θέματα εξακολουθεί να είναι δύσκολη, αν και χαιρετίζουμε τις συστάσεις ε, της, ανεξάρτητης, της έκθεσης της Ανεξάρτητης Επιτροπής Έρευνας του Μπαχρέιν. Αναφέρθηκα στο, κατεπήγον, στο ψήφισμα κατεπήγοντος του Ιανουαρίου. Η αντιπροσωπεία που πήγε στο Μπαχρέιν, λοιπόν, πιστεύω ότι ήταν πολύ καλά προετοιμασμένη για να συζητήσει τα πολλά και διάφορα θέματα. Και τώρα δίνω το λόγο στην κυρία Μπαϊτιέρε, που είναι πρόεδρος της αντιπρο... ήταν πρόεδρος της αντιπροσωπείας και να μας κάνει την ενημέρωση. Ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγικά σας σχόλια. Όπως ακούσατε ήδη, υλοποίησαμε την ε, αποστολή στον Μπαχρέιν, στείλαμε την αντιπροσωπεία και να ρωτήσω, έχεις φέρει την έκθεση, είναι έτοιμη έκθεση. Ζεστή είναι η έκθεση ακόμη. Έκανα τις τελευταίες διορθώσεις χθε το βράδυ και τώρα είναι έτοιμη η έκθεση. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό το σχέδιο της έκθεσης ε, το λάβαμε το Σαββατοκύριακο, την περασμένη εβδομάδα. Εγώ και οι συνάδελφοι από την Εντροπροσωπεία εργαστήκαμε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού για να προετοιμάσουμε την τελική εκδοχή του σχεδίου τους έκθεσης. Ο κύριος Χάουιτ ε, υποσχέθηκε ότι σήμερα θα παρευρεθεί εδώ μαζί μας, ελπίζω να έρθει σύντομα. Αλλά θα αρχίσω να ενημερώνω για την επίσκεψή μας. Αναφέρεται το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κατεπήγοντα. Πρέπει να ομολογήσω ότι δεν ήμουν ιδιαίτερα υπέρ αυτού γιατί νόμιζα ότι καταρχήν έπρεπε να συζητήσουμε τη δική μας έκθεση. Γιατί πήγε και η αντιπροσωπεία τόπου είδαμε λοιπόν τα πράγματα από μέσα και... Αν θέταμε το ψήφισμα λίγο αργότερα, αφού θα είχε συζητηθεί αυτή η έκθεση, νομίζω ότι θα ήταν πιο παραγωγική διαδικασία. Κατά την άποψή μου, το ψήφισμα δεν ήταν τόσο ισορροπημένο όσο θα ήθελα. Αλλά να τονίσω ότι ο πρωταρχικός στόχος της αποστολής μας ήταν ε, να αξιολογήσουμε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον Μπαχρέιν. Όπως ξέρετε, στον Μπαχρέιν είχαμε μια μακρά περίοδο διαδηλώσεων που ξέσπασαν νωρίς το 2011 και είχαμε καταστολή από την πλευρά της κυβέρνησης ε, με πράξεις βίας και ορισμένες ε, δράσεις εξακολουθούν ε, να λαμβάνουν χώρα, εξακολουθούν να υποφέρουν οι άνθρωποι, αλλά η κατάσταση στα δικά μου μάτια και στα μάτια της αντιπροσωπείας σε μεγάλο βαθμό είχε σταθεροποιηθεί. Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν μαζικές διαμαρτυρίες, ε, υπάρχει μαζική βία στο δρόμο, αλλά Φυσικά υπάρχουν ορισμένα περιστατικά. Θα σας ενημερώσω εν συντομία για τις συναντήσεις μας. Μπορέσαμε να συναντηθούμε με ιδιαίτερα υψηλού ε, εκπροσώπους της κυβέρνησης, τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Υπουργό Δικαιοσύνη, τον Υπουργό Εξωτερικών μας ε, συνόδευε ο Αμπτούλη Ραχμάν Ρατσίτ Μουμπάη, ο οποίος είναι επικεφαλής ε, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και πρέπει να ευχαριστήσω και τον κύριο Κούλακ, ο οποίος είναι ο πρεσβευτής μας. Ομαλά διεξήθηκε το έργο της αντιπροσωπείας ε, και πραγματικά εκπληρώθηκαν οι επιθυμίες μας να συναντήσουμε κάποια πρόσωπα. Θα σας αναφέρω και την επισκέψη μας στη φυλακή που οργανώθηκε επί τόπου. Και νομίζω ότι πρέπει να αναφερθεί. Επίσης, συναντηθήκαμε με εκπροσώπους της αντιπολίτευσης, εκπροσώπους ε, του τύπου, υπερασπίστες των ανθρωπινών δικαιωμάτων, του κινήματος της αντιπολίτευσης και άλλους. Μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες στην εκθεσή μας. Στην έκθεσή μας επίσης αναφερθήκαμε θίγουμε μάλλον το πώς βλέπουν τα πράγματα οι πρεσβευτές από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επίσης ε, θέλουμε να κατανοήσουμε πόσο μακριά οι συστάσεις ε, της Ανεξάρτητης Εξεταστικής Επιτροπής ε, του Μπαχρέιν ήταν ανεξάρτητες. Ρωτούσαμε κάθε φορά σε ποιο βαθμό πληρούνται ή έχουν ικανοποιηθεί οι συστάσεις αυτές. Πάντως αυτές οι συστάσεις ήδη εφαρμόζονται σε μεγάλο βαθμό. Αλλά φυσικά θέλαμε να δούμε και πού θα ήταν η προθεσμία πότε θα υπάρξει αυτή η εφαρμογή. Επίσης, οι πρεσβευτές τόνισαν ότι είναι πολύ συντηρητική η αντιπολίτευση ενίοτε και η κυβέρνηση βλέπει και άμεση παρέμβαση του Ιράν μέσω της μειονότητας των Σιητών στις κρατικές υποθέσεις. Επομένως, Τονίστηκε σε πολλές από τις συναντήσεις μας ε, το θέμα των σχέσεων με τις άλλες χώρες. Ως ένα θετικό βήμα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι έχουμε το Διεθνές Ίδρυμα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Συναντήσαμε τον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος μας είπε ότι δύο χρόνια υπάρχει αυτή η Επιτροπή και υπήρξαν 28 ε, δηλώσεις που δημοσιεύτηκαν κατά της κυβέρνησης και 300 περιπτώσεις παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων που περιλαμβάνονταν στην ετήσια έκθεση. Αυτό το βήμα θα μπορούσε να θεωρηθεί ως θετικό, όμως ο Γενικός Γραμματέας τόνισε επίσης ότι οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες περιορίζονται επειδή συνεχίζονται εσωτερική σύραξη. θα ήθελα να φέρω τα πιο πρόσφατα νέα. Θέλει τώρα ο Βασιλιάς ε, να ξεκινήσει το διάλογο και η αντιπολίτευση ε, δηλώνει ικανοποίηση από την πρόθεση αυτή του Βασιλιά. Και η κοινωνία να έχει κάποιες συνεισφορά σε αυτήν την πολύ θετική απόφαση και εμεί διαδραματίσαμε ένα ρόλο σε αυτήν την πολυθετική απόφαση, γιατί αυτό ζητήσαμε. Επίση, συναντηθήκαμε πολλάκι, ε, μάλλον είχαμε πολλέ συναντήσει με εκπροσώπου του κατώτερου αλλά και του, του κάτω και του άνω κοινοβουλίου. Και μπορώ να σας πω ότι με εξέπληξαν ε, πόσο επικριτικοί είναι οι βουλευτές για την κατάσταση και για το τι έχει γίνει. Όμως ε, ήταν κάπως όφρονες στις παρατηρήσεις τους για πιθανές μεταρρυθμίσεις στο μέλλον. Ήταν νομίζω πολύ παραγωγικές αυτές οι συζητήσεις και τονίσαμε ότι οι επόμενες κοινοβουλευτικές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για το 2014 Πρέπει να προετοιμαστούν οι κανόνες ε, γέρος ε, και θα πρέπει να υπάρχουν στοιχεία εθνικής συμφιλίωσης. Ρωτήσαμε, γιατί αυτή η σύσταση ανεξάρτητης επιτροπής δεν έχει λάβει ακόμη χώρα. Οι συνομιλητές μας μας είπαν ότι δεν είναι τόσο σταθερή η κατάσταση προκειμένου να εφαρμοστεί αυτή η σύσταση τώρα έχουν σκοπό να την εφαρμόσουν στο μέλλον. Αλλά τώρα είναι κάπως πιο προσεκτική απέναντι στην εφαρμογή όλων των συστάσεων. Συνολικά θα έλεγα ότι εμείς οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι βουλευτές του Μπαχρέιν ε, συμφωνήσαμε σε μια επικοδομητική συνεργασία μεταξύ μας για τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα και ευημερία της χώρας. μιλήσαμε, συζητήσαμε το θέμα της άσκησης υπερβολικής βίας από την πλευρά της αστυνομίας. Και σε μια συζήτηση με τον Υπουργό Εσωτερικών, ανέφερα ότι έχουν ερευνηθεί ήδη κάποιες υποθέσεις και έχουν τιμωρηθεί ένοχοι. Επίσης ρωτήσαμε τι γίνεται με τους απολυμμένους εργαζομένους κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών. Πολλοί δεν πήγαν στη δουλειά τους και στις περισσότερες περιπτώσεις σε οκτώ περιπτώσεις είχαν επιστρέψει αυτοί οι εργαζόμενοι αλλά εξακολουθούσαν να υπάρχουν δυσκολίε με, τον ιδιωτικό, με τον ιδιωτικό τομέα. Στο δημόσιο φαίνεται ότι είχε επιληθεί το ζήτημα αυτό επιστροφή στι εργασίε του. Επίσης, μιλήσαμε για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την κοινωνία των πολιτών. Συζητήσαμε και με άτομα, ως άτομα και ως αντιπροσωπεία. Επίσης, δημοσιεύσαμε μία δήλωση στον τύπο, όπου τονίσαμε ότι πολλά πρέπει να γίνουν ακόμη για να διασφαλίσουμε πραγματική ελευθερία των μέσων και υπογραμμίσαμε τη σημασία του πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης καθώς και την ανάγκη ελεύθερης έκφρασης για τα κοινωνικά μέσα και απευθύναμε έκκληση να μπορούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση δημοσιογράφοι στη χώρα. Είχε δημοσιευτεί ένα άρθρο πριν την επίσκεψή μας και ρώτησα γιατί δεν επιτράπει το δημοσιογράφο να μπει στη χώρα. Και η απάντηση που πήρα ήταν η εξή. Ότι δεν απέκτησε τη σωστή θεώρηση. Ήταν ε, λάθος η θεώρηση που είχε δει ο δημοσιογράφος και έτσι δεν του επέτρεψε να μπει στη χώρα. Αυτή την απάντηση λάβαμε. Και ο Ρίτσαρτ ε, ήταν μπροστά όταν θέσαμε την ερώτηση για ένα βουλευτή που δεν ε, πήρε τη θεώρηση. Μας απάντησαν ότι δεν έφτανε ο χρόνος να προετοιμαστεί τη θεώρηση για το μέλος της αντιπροσωπείας μας. Σύμφωνα με την ε, πλευρά του Μπαχρέιν, δεν παρουσιάστηκαν τα έγγραφα στην πρεσβεία του Μπαχρέιν έγκαιρος. Γι' αυτό και ο συνάδελφος δεν έλαβε τη θεώρηση. Νομίζω ότι πολύπλοκη είναι η υπόθεση των γιατρών. Γιατί συζητήσαμε και με την αντιπολίτευση αλλά και με τους γιατρούς στο Μπαχρέιν και δηλώσαμε στον τύπο ότι είμαστε αντίθετοι στην κατάσταση το ιατρικό προσωπικό να υπόκειται σε δικαστική παρενόχληση και σε φυλάκιση μόνο επειδή ασκεί το λειτουργήμά του. Δηλώνεται σαφώς. Όμως, οι εκπρόσωποι του ιατρικού κλάδου του Μπαχραήν μας είπαν ότι αυτές οι φυλακίσεις και επαγγελίες κατηγοριών δεν είχαν να κάνουν με, το, με τα καθήκοντά τους, με την επιτέλεση των καθηκόντων τους, αλλά επειδή δεν προσέφεραν ε, θεραπεία σε κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους και χρησιμοποίησαν τις εγκαταστάσεις ε, του ιατρικού ίδρου Αλμάνια για κάποιες άλλες διαδικασίες πέραν ε, της θεραπείας. Αλλά ο μόνο τρόπο να λυθεί αυτό το πρόβλημα θα είναι να είναι ανοιχτή και δίκαιη η δίκη. Συζητήσαμε αυτό το θέμα όταν συναντηθήκαμε με τον Υπουργό Δικαιοσύνη και τον Υπουργό Εσωτερικών. Ο Υπουργό Δικαιοσύνη αναγνώρισε ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, πολλές υποθέσεις που πρέπει να συζητηθούν και να επιληθούν. Και επίσης, τόνισε ότι υπάρχουν πολλοί δικαστές δεν είναι αρμόδιοι. Δεν έχουν τα κατάλληλα προσόντα να κάνουν τη δουλειά τους. Και πρέπει να βελτιωθούν τα προσόντα τους. Και καλώ όρισε την πρότασή μας να βοηθήσουμε εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση να εκπαιδεύσουμε τους δικαστές. Και να δημιουργήσουμε ένα σύστημα που να διασφαλίζει την υλοποίηση δικής δίκης, την εξαγωγή δικής δίκης. Ως κάτι θετικό μπορούμε να τονίσουμε ότι έχει ε, διοριστεί και ο συνήγορος του πολίτη Όμως, νομίζουμε ότι τα δικαστήρια θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα και όλοι οι οργανισμοί που ασχολούνται με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως και ο Σύνολο του Πολίτη, θα πρέπει να είναι ανεξάρτητε. Και υπάρχει αυτό και στην δήλωσή μας στον τύπο. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, γιατί είναι εδώ και ο κύριο Χάουιτ. Και θα προσθέσει κάποιες πληροφορίες. Θα λέγω ότι πολλά ήδη έχουν γίνει. Θέλουμε το σχάρι. Συνήγορο του πολίτη που ανέφερα και το ότι η δικαστική εξουσία έχει διαχωριστεί. Έχει ξεκινήσει ο διαχωρισμός ε, του δικαστικού σώματος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Δεν έχει ολοκληρωθεί βέβαια ακόμα και έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες ε, για να υπάρξει ελευθερία της έκρασης υποστήριξη των δικαστικών ερχών, προστασία των θυμάτων και άλλες συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσει προκειμένου να ενισχυθεί ο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Νομίζω ότι λάβαμε και μια θετική πληροφορία μετά την επίσκεψη ότι σε κάποια αστυνομικά τμήματα ήδη υπάρχει εξοπλισμός οπτικοακουστικός για να αποφεύγεται, να αποφεύγονται τα βασανιστήρια των κρατουμένων. Ακούσαμε ότι βασανίζονται οι άνθρωποι. Και βέβαια αυτό μας λύπησε. Και όπως είπα, αυτή η επίσκεψη στη φυλακή οργανώθηκε με επιχειρησιακό τρόπο το πρωί. Το ζητήσαμε από τον Υπουργό Δικαιοσύνη και κατόπιν συναντηθήκαμε και με τον Υπουργό Εσωτερικών και πραγματικά μας επέτρεψε να πάμε στη φυλακή. Ζητήσαμε να περάσουμε μια μισή ώρα ε, στη φυλακή μαζί με ανθρώπους που υπερασπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά τελικά παραμείναμε εκεί πολύ περισσότερο. Και το εκτιμήσαμε αυτό, γιατί δεν μπορώ να είμαι σίγουρο ότι σε πολλές χώρες θα μας επέτρεπαν κάτι τέτοιο. Γιατί μια φυλακή είναι μια φυλακή. Αλλά πράγματι μπορούσαμε να μιλήσουμε απευθεία, ένα προ ένα με τους φυλακισμένους. Ε. Έτσι λοιπόν μπορούσαμε να δούμε τα πράγματα από μέσα. The report is... Η έκθεση αποτελείται από 15 σελίδες, είναι μακροσκελής. Προσπάθησαμε να είμαστε όσο δυνατόν πιο αντικειμενικοί για να συζητήσουμε την κατάσταση από διάφορες οπτικές και νομίζω ότι και η, η δήλωση στον τύπο ήταν επικριτική, μεν, αλλά ενθαρρύνει δε να γίνουν κάποια θετικά βήματα. Νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε το διάλογο με τους βουλευτές του Μπαχρέιν και με την κυβέρνηση. Ως επικεφαλής της αντιπροσωπείας με διαβέωσαν πολλές φορές ότι η κυβέρνηση του Μπαχρέιν επιθυμεί να συνεχίσει το διάλογο μεταξύ των ε, ομάδων των διαφορών συνομιλητών. Και θέλω να σας αναφέρω ότι είπε ο Εσωτερικών. Είπε ότι όλοι οι Σουνίτες οι ε, είναι πολίτες του Μπαχρέιν. Δεν θα θέλαμε να κάνουμε διακρίσεις. εξακολουθεί να μην είναι δυνατό ένα τμήμα του πληθυσμού να μπορεί να συμμετέχει στις δυνάμεις ασφαλείας, αλλά μπορούν να είναι στο στρατό. Νομίζω ότι με την εμπειρογνωμοσύνη μας ε, μπορούμε να συμβάλλουμε για βελτίωση της κατάστασης στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την εξαιρετικά λεπτομερή έκθεση. Ο κύριος Χάουαρτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τη συνάδελφο η οποία ηγήθηκε της αποστολής μας και θα ήθελα να την ευχαριστήσω για αυτό το δύσκολο έργο που ανέλαβε και μπορώ να πω ότι η περιγραφή που σας έδωσε της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον Παχρέιν ήταν πλήρης και δίκαιη. Γι' αυτό εγώ θα ήθελα απλώς να προσθέσω ορισμένα στοιχεία. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Γραμματεία γνωρίζετε ότι κατά το παρελθόν είχα ασκήσει κάποια κριτική. Γιατί θεωρώ ότι θα, θα πρέπει να δώσουμε το, τη, φωνή στα θύματα των, παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τις επισκέψεις μας σε χώρες και θεωρώ ότι σε αυτή την επίσκεψη το καταφέραμε να το κάνουμε αυτό και πιστεύω ότι η υποστήριξη που είχαμε από τις Βρυξέλλες προς αυτή την κατεύθυνση και αυτή την προσπάθεια ήταν σημαντική γιατί εξάλλου η διοργάνωση της αποστολής αυτής ήταν δύσκολη και θέλω να σας ευχαριστήσω και να καταγραφεί, να ζητήσω να καταγραφεί αυτό και στα πρακτικά. Και να ε, θεωρώ ότι πρέπει να συγχαίρουμε εκείνους που εργάζονται σκληρά όταν το καταφέρουν. Λοιπόν, επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον πρέσβη μας, τον αντιπρόσωπό μας, για τις, και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, αλλά και για τις επαφές που είχαμε μετά την αποστολή. είχαμε σημαντική συνεργασία και αυτό βοήθησε την διεξαγωγή της αποστολής μας εκεί. Βεβαίως συζητήσαμε πολλά ζητήματα με την κυβέρνηση του Μπαχρέιν με στόχο την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με στόχο να διαπιστώσουμε την κατάσταση και να κάνουμε κάποιες προτάσεις και κάποιες παρατηρήσεις. Θεωρώ ότι και δικιά της την πλευρά η κυβέρνηση του Μπαχρέιν θα θεωρούσε την επίσκεψή μας επιτυχημένη στα ζητήματα της ελευθερίας της έκφρασης. Το Μπαχρέιν παραμένει μια χώρα στην οποία αν κάποιο ασκήσει κριτική στην βασιλική οικογένεια θα μπει στη φυλακή. Και αυτό είναι καταγεγραμμένο στο δίκαιο του, στο, στην νομοθεσία. Άρα είναι σαφές ότι η ελευθερία της έκφρασης στο Μπαχρέιν είναι προβληματική, καθώς επίσης και η ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωση, Γι' αυτό και τα κοινωνικά μέσα δικτύασης έχουν αποκτήσει τόσο μεγάλη σημασία και έχουν γίνει τόσο δημοφιλή Έχουμε δει πολλές, πολλούς ανθρώπους να συλλαμβάνονται εξαιτίας απόψεων που εξέφρασαν σε κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Άρα, στην συζήτηση που είχαμε με τους εκπροσώπους του Μπαχρέιν, διαπιστώνουμε τη διαφορά για παράδειγμα, στη χώρα μου, αν κάποιο θέλει να εκφραστεί κατά τη βασιλική οικογένεια, γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να μην αρέσουν σε κάποιον, έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Στον Παχρέν δεν ισχύει αυτό. Σε σχέση με του κρατουμένου συνείδηση. Ποτέ δεν καταφέραμε να διαπιστώσουμε τον ακριβή αριθμό των κρατουμένων συνείδηση. Έχουμε διάφορε εκθέσει που λάβαμε πριν την επίσκεψή μα. Ακούμε για χιλιάδε κρατουμένου συνείδηση, τρει χιλιάδε πιθανόν. Ορισμένοι από αυτού είχαν κρατηθεί προσωρινώ και το ερώτημα παραμένει πόσοι από αυτού παραμένουν στη φυλακή. Δεν καταφέραμε να το διαλευκάνουμε παρόλο που ζητήσαμε επανειλημμένα συγκεκριμένα στοιχεία. Αυτό είναι επίση ένα ζήτημα που μα ανησυχεί. Η απελευθέρωση των κρατουμένων συνείδηση θα ήταν ένα σημαντικό βήμα που θα μπορούσε να λάβει η κυβέρνηση του Μπαχρέιν για να προωθήσει το διάλογο και να οικοδομήσει εμπιστοσύνη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν κρατούμενοι συνείδησης οι οποίοι έκαναν έφεση και απερίφθη η έφεσή τους και παραμένουν στην φυλακή και προφανώς οι περιπτώσεις αυτές έχουν εμβληματική σημασία. Θα ήθελα να επισημάνω λοιπόν το ζήτημα αυτό των κρατουμένων συνείδηση στην Επιτροπή μας. Τώρα σε σχέση με την Ανεξάρτητη Εξεταστική Επιτροπή υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Διαφορετικά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν διαφορετικές απόψεις. Το 25% των προτάσεων αυτής της Επιτροπής κατά την κυβέρνηση έχουν ε, εφαρμοστεί θεωρούμε αλλά ενώ η κυβέρνηση του Μπαχρέιν μας λέει ότι το 98% των συστάσεων εφαρμόστηκαν, άρα μπορούμε να συνεχίσουμε να διαφωνούμε, μπορούμε να συνεχίσουμε να διαφωνούμε και με τους συνομιλητές μας στο Μπαχρέιν, αλλά νομίζω όλοι θα συμφωνήσουμε ότι η υλοποίηση των συστάσεων της Ανεξάρτητης Εξεταστικής Επιτροπής θα ήταν ένα σημαντικό βήμα πρόοδου. Ε, προσωπικά αμφιβάλλω σοβαρά κατά πόσον έχουν εφαρμοστεί στη πράξη αυτές οι συστάσει. Τώρα στη σχέση με τους εκπαιδευτικού, όπως επίσης και με τους ιατρούς, στο οποίο αναφερθήκατε πριν. Συναντηθήκαμε με αρκετού, που μας είπαν ότι είτε είχαν φυλακιστεί στο παρελθόν είτε αναμένουν να παραπεμφθούν σε δίκη. Για παράδειγμα, στην περίπτωση των ιατρών επειδή είχαν περιθάλψει Διαδηλωτέ και έτσι είχαν περιέλθει στην κατοχή τους ε, αποδεικτικά στοιχεία που επιδείκνυαν βασανιστήρια. Αυτά, αυτές οι περιπτώσεις, σαφέστατα είναι περιπτώσεις που είχαν την διεθνή ε, προσοχή, την προσοχή της διεθνούς κοινή γνώμης, αλλά υπάρχουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι είτε μπήκαν στη φυλακή, είτε απειλήθηκαν με παραπομπή στη δίκη με φυλάκιση, είτε έχασαν τη δουλειά τους σε τέτοιου είδους καταστάσεις και για τους οποίους δεν δημοσιοποιήθηκαν τόσο τα στοιχεία. Στο ζήτημα της κακομεταχείρισης και των βασανιστήριων, το Υπουργείο Εσωτερικών μας είπε ότι χρησιμοποιήθηκαν πραγματικές σφαίρες κατά διαδηλωτών, χωρίς να λάβει θέση για το κατά πόσο οι διαδηλωτές αυτή την ειρηνική, αλλά ε, το θέσαμε το ζήτημα ενώπιον του, των συνομιλητών μας από τον ένα ζήτημα που μας είχαν ετέθη από οργανώσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για πυροβολισμούς σε απόσταση με ε, πλαστικές σφαίρες αλλά σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου πράγμα που τις καθιστά θανατηφόρες. Καθώς επίσης και χρήση δακρυγόνων. Τύπου τοπικέ οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν πει ότι πιθανώς τα χημικά, στη χημική σύνθεση των δακρυγόνων που χρησιμοποιούνται στον Παχρέιν να μην ε, είναι μια χημική σύνθεση που θα ήταν αποδεκτή στις ευρωπαϊκές χώρες. Μπορούμε με όλα αυτά τα περιστατικά να συμπεράνουμε ότι η ελευθερία του συναθρίζεστε δεν γίνεται σεβαστή. Τώρα, κάποιε παρατηρήσει για τον ίδιο το διάλογο και με αυτέ θα κλείσω. Προφανώ και ζητήσαμε να συνεχιστεί ο διάλογο, γιατί είναι ο μόνο τρόπο να προχωρήσουμε και πράγματι το Μπαχρέιν αυτό επιθυμεί. Και θεωρώ ότι ε, αυτό είναι και το σωστό, αυτό πρέπει να κάνουμε. Δεν έχει νόημα να απλώ να καταγγέλουμε και να πούμε ότι μια πλευρά έχει δίκιο 100% ή άδικο 100%. Να συνεχίσουμε λοιπόν το διάλογο με όλες, όλα τα μέρη της κοινωνίας. Αλλά από τη στιγμή που το λέμε αυτό και από τη στιγμή που θέλουμε να, να γίνει ένας πραγματικός διάλογος που να τον εμπιστεύονται τα μέρη που συμμετέχουν σε αυτόν, δεν μπορώ παρά να μην διαπιστώσω ότι βρισκόμαστε πολύ μακριά από μια τέτοια κατάσταση. Δηλαδή είναι ένα πράγμα η κυβέρνηση να λέει ότι επιθυμεί το διάλογο και είναι άλλο πράγμα να δημιουργήσει τι συνθήκε εντό των οποίων να μπορεί να διεξαχθεί πραγματικά ένα τέτοιο διάλογο. Τώρα, πιστεύω ότι θα είναι ενδιαφέρον να διαβάσετε την αναφορά που μόλις σας μοιράστηκε. Αλλά θα ήθελα να σας επισημάνω ότι μέρη της αντιπολίτευσης δεν συμμετέχουν στον διάλογο. Και δεν θα πρέπει να αποκλειστεί κανείς από αυτό το διάλογο. Πρέπει να είναι πλήρως πλήρης η συμμετοχή. Έχει συμφωνήσει η κυβέρνηση του Μπαχρέιν επ' αυτού και είναι μια χώρα που είναι πιο ανοιχτή σε ορισμένους, προς ορισμένες ομάδες, προς, ορισμέν, στην περιοχή, χωρίς αυτό προφανώς ποτέ να είναι α, δικαιολογία. Ας μην ξεχνάμε ότι άλλες περιοχές στην περιοχή του Περσικού κόλπου είναι λιγότερο ανοιχτές. Άρα το γεγονό ότι διαπιστώνουμε τόσε παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν σημαίνει ότι το Μπαχρέιν είναι σε χειρότερη κατάσταση από ότι άλλοι γειτονέ του αλλά είναι μια χώρα στην οποία χρειάζονται μεταρρυθμίσεις, δεν ε, έχουν υπάρξει τα αποτελέσματα ας πούμε, της Αραβικής Άνοιξης ακόμα δεν είναι ορατά, αλλά παραμένουν σημαντικές και σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είναι και ένας από τους λόγους που η Επιτροπή, που η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποφάσισε κατά προτεραιότητα να επισκεφθεί την χώρα. Ελπίζω η επίσκεψή μας να βοήθησε να βελτιωθεί η κατάσταση στον Παχρέν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ρίτσαρτ Χάουιτε, για την ενημέρωση. Η κυρία Αντρικένη και η κυρία Σίνκλερ είναι δύο νέα μέλη. Ήθελαν και εκείνες να μιλήσουν, αλλά είναι σε αποστολή στη Χιλή. Οπότε ζήτησαν να αναβληθεί η έκθεση. Αυτό δεν γινόταν. Τους παρέπεμψα σε μια συνάντηση με την ΑΦΕΤ που θα γίνει στις 7 Μαρτίου. Εκεί οι θα ε, υπάρχουν τα μέλη της αντιπροσωπείας του Μπαχρέιν. Ο πρέσβης ε, θέλει να λάβει το λόγο. Κύριε πρέσβη, θα διευκολύνετε τη δουλειά μου αν περιοριστείτε σε ένα τρίλεπτο. Αυτό είναι ο γενικός κανόνας εδώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Βάιντερα και την αντιπροσωπεία που πήγε στο Μπαχρέιν και που έκανε αυτή την έκθεση. Δεν θα σχολιάσω την έκθεση, αλλά αυτή είναι η έκθεση της επίσκεψης. Εμείς θέλαμε την επίσκεψη για να ανοίξουμε διάβλους επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης του Μπαχρέιν για να απαντήσω στον κύριο Χάουιτ για τον εθνικό διάλογο. Πριν από λίγες μέρες ε, ε, ο ε, μεγαλειότητα του, ο βασιλιάς, ζήτησε διάλογο και τώρα ετοιμαζόμαστε για αυτό τον εθνικό διάλογο που θα λάβει η χώρα σύντομα. Όπως είπα, θέλαμε να γίνει επίσκεψη για να δείξουμε την καλή μας θέληση και την καλή συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών. Τώρα σκέφτομαι δυνατά. Από την περασμένη εβδομάδα διαρωτώμην τι έγινε. Η λογική λέει ε, υπάρχουν κάποια βήματα. Το ένα είναι ότι έγινε η επίσκεψη, το 2 η έκθεση, το 3 τα συμπεράσματα. Όμως στις 17 Ιανουαρίου την περασμένη εβδομάδα εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο ένα ψήφισμα κατά του Μπαχρέιν και σκέφτομαι δυνατά τώρα γιατί δηλαδή σπεύσαμε να βγάλουμε αυτό το συμπέρασμα. Η μόνη εξήγηση είναι ότι υπάρχουν ορισμένα μεγέθη κρίσιμα ή μάλλον προσωπικότητες κρίσιμες και κέρυες που στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο δεν θέλουν να ανοίξει αυτή η πόρτα της συνεργασίας. Και ε, έτρεξαν, ε, έσπευσαν να κλείσουν την πόρτα. Πιστεύω όμως ότι θα παραμείνει ανοιχτή και όλοι είστε ευπρόσδεκτοι. Επίσης κάθε φορά σκέφτομαι που θα γίνεται επίσκεψη στον Μπαχρέιν, θα ακολουθεί ψήφισμα κατά της χώρας μου. Ελπίζω όχι, γιατί δεν θα βοηθήσει κάτι τέτοιο. Η Επιτροπή θα μπορούσε ίσως ε, να κάνει μια τελική δήλωση σχετικά με την επίσκεψη, δηλαδή αναφέροντας κάποια θετικά, ευχαριστώντας την κυβέρνηση, γιατί περασμένη εβδομάδα είχαμε το ψήφισμα και σκέφτομαι και το υποβάλλω αυτό και στην Πρόεδρο και στην Επιτροπή ε, ως πρόταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρέσβη, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν ε, σχεδιάζουμε να γίνουν μαζί επισκέψεις και ψηφίσματα. Αυτά τα ψηφίσματα για τα κατεπήγοντα έχουν άλλη λογική και αναφέρονται σε θέματα που αφορούν τη χώρα, καταστάσεις που λαμβάνουν χώρα εκεί. Πρέπει όμως να δούμε και τη διαδικασία του κατεπήγοντος Και τώρα έχουμε συναδέλφους, την κυρία Στάντε από την ΙΑΕΣΕ, από την Αραβική Χερσόνησο και τον κύριο Αντώνη Αλεξανδρίδη από τη Μονάδα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να μας πείτε ε, σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα κατεπήγοντος που εγκρίναμε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν να εκφράσω την αναγνώρισή μας του ρόλου που παίζει το Κοινοβούλιο για να φροντίσει ότι η κατάσταση στο Μπαχρέιν θα παραμείνει στην δημόσια ανοιχτή ατζέντα. Να ευχαριστήσω επίσης για την συμβολή της Υποεπιτροπής και τις πολύ ισορροπημένες συστάσεις και εκθέσεις. Ε, είναι πολύ σημαντικό θέμα για την ύπατη εκπρόσωπο η κατάσταση εκεί, γιατί η ε, ευημαϊρία των κατοίκων του Μπαχρέν και η αποφυγή βίας από όλες τις πλευρές βρίσκεται στο επίκεντρο των δράσεων που αναλαμβάνει. Ο εθνικός διάλογος όμως πρέπει να γίνει πιο στιβαρός, στέρεος Χαιρόμεθα για την ε, έκκληση που απέθυνε ο Βασιλέας για νέο γύρο εθνικού διαλόγου μετά από μια έκκληση και του πρίγκιπα και δόθηκε και από την αντιπολίτευση μια ενθαρρυντική απάντηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχώς ζητούσε από όλα τα μέρη να προετοιμάσουν το έδαφος για έναν εθνικό διάλογο, για βιώσιμες μεταρρυθμίσεις ε, ε, ασχολούμενοι επίσης και με τις δυσκολίες σε οικονομικό επίπεδο του λαού του Μπαχρέιν. Αναφερόμενοι σε ένα θέμα που έθεσε το αξιότιμο μέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση πράγματι τώρα δημιουργεί ένα πρόγραμμα το οποίο εστιάζει κυρίως στις ε, συστάσεις της Επιτροπής Πατσιούνη για την εκπαίδευση δικαστών και εισαγγελέων. Τώρα το καταρτίζουμε αυτό το πρόγραμμα. Να πω επίσης ότι η Πατή Εκπρόσωπος εξέφρασε απογοήτευση για την απόφαση να μην υπάρξουν για τις ποινές νωρίτερα το μήνα, γιατί θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει επιοίκεια ε, σε αυτές τις καταστάσεις, σε αυτές τις περιπτώσεις. Εσείς δεν θα προσθέσετε τίποτε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τάνοκ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συγγνώμη που δεν ήμουν στην αρχή της συζήτησης και δεν ήμουν στην αντιπροσωπή, αλλά συμμετείχα στο ψήφισμα στο Στρασβούργο και συζητήσει στην Ολομέλεια. Να κάνω μερικά σχόλια σχετικά με το βασίλειο του Μπαχρέιν. Είναι μικρή χώρα που αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις. Προσπαθεί να διατηρήσει τη συνταγματική μοναρχία και την ανεκτική πολυεθνική κοινωνία με πολλές θρησκείες. Το Ιράν θα ήθελε Ισλαμική δημοκρατία με νόμο Συρίας, ε, ε, Σαρίας. Ε, υπάρχουν τέτοιες προσπάθειες. Ε, ο βασιλιάς και η κυβέρνηση αναγνωρίζουν τα λάθη, ε, δυσανάλογη χρήση δύναμης πριν από ένα χρόνο ενάντια στους διαδηλωτές και ακολουθήθηκε σωστή διαδικασία για να αντιμετωπιστούν αυτά. Εις ό,τι αφορά την, τις ποινές που επιβλήθηκαν, ζητήσαμε επί οίκια ε, σε σχέση με ορισμένε ε, αποφάσεις. Αναμφίβολα το Μπαχρέιν πρέπει να μάθει περισσότερα πράγματα σχετικά με το πώς θα εφαρμόζει τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, με δημοκρατικό τρόπο και εκείνοι αναγνωρίζουν ότι δεν είναι η τέλεια δημοκρατία αλλά με βάση τα πρότυπα της περιοχής είναι πάρα πολύ ανεκτική η χώρα έχουν χριστιανικές εκκλησίες έχουν μεγάλη ανεκτικότητα απέναντι σε άλλες θρησκείες και νομίζω ότι θα ήταν δυσανάλογο να εστιάσουμε εκεί. Είναι μια πολύ μεγαλύτερη χώρα στην περιοχή που είναι πολύ επιθετικότερη και δυσάρεστη σχετικά με την αντιμετώπιση των μειονοτήτων. Το Μπαχρέιν μαζί με τα Εμμυράτα προσπαθεί να ε, διατηρήσει την ασφάλεια και την ακαιρεότητα στη χώρα και να απομακρύνει το ενδεχόμενο ξένης ε, επέμβασης. Πολλές φορές αντιμετωπίζουμε διλήμματα με τα ανθρώπινα δικαιώματα για να εξισορροπήσουμε καταστάσεις και θα ήταν άδικο ιδιαίτερα αν θεωρεί ο πρέσβης εδώ ότι στοχοποιείται και από ένα ψήφισμα που είναι αρκετά επικριτικό και από μια συζήτηση εδώ στην Υποεπίτροπη που ε, βάζει στο στόχαστρο το Μπαχρέιν και το αναδεικνύει και το απομονώνει για να τονίσει υπερβολές ή σοβαρές καταχρήσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα. Έγιναν λάθη και η κυβέρνηση νομίζω τα αναγνωρίζει και θα αντιδράσουν στα αιτήματα τα δικά μας για βελτιώσεις και για επανεξέταση αυτών των υποθέσεων και ίσως ο βασιλιάς θα δείξει και όπου χρειάζεται. Ευχαριστώ κύριε Τάνοκ. Και σωστά αναφέρατε το τι ισχύει στην περιοχή και είπα στην αρχή ότι ο Υπουργό Δικαιοσύνη τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε την επίσκεψη και νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε μαζί του τι παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κύριε Πρεσβευτά, εσεί ρωτήσατε αν υπάρχει κάποια τελική δήλωση που θα προκύψει από εδώ. Η τελική έκθεση της αντιπροσωπείας ε, που μόλις τυπώθηκε νομίζω ότι θα δώσει μια πολύ λεπτομερή εικόνα των πορισμάτων και αυτή είναι η τελική δήλωση. Επίσης, ε, ξέρετε ότι ό,τι συζητάμε εδώ αναμεταδίδεται ζωντανά στο διαδίκτυο και μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε όλες τις δηλώσεις και το έγγραφο. Σας ευχαριστώ και πάλι όλους ε, για τα σχόλια. Λοιπόν, έχω δύο άτομα που ζητούν το λόγο. Να πω δύο λόγια, κυρία Βάιντερα. Ρίτσαρ, θες εσύ πρώτο το λόγο. Μπορεί να τα έλεγε και εσύ αυτά. Αλλά μπορεί να δείξει η έκθεση ότι έχει δίκιο ο κύριος Τάνοκ. Σα θέλω να απαντήσω στο πρεσβευτή. Εγώ δεν θα είχα αντίρρηση αν ε, η αντιπροσωπεία εξέφραζαν τις ευχαριστίες μας στον Παχρέιν για τη φιλοξενία τους. Το έκαναν αυτό, δεν ξέρω αν αυτό τώρα παραβιάζει ε, ουσιαστικά το λειτουργήμα μας, ε, αλλά ίσως θα έστειλε ένα μήνυμα, αν το πράταμε. Και ανυπομονώ να συναντηθώ με τους βουλευτές, ε, του Μπαχρέιν ε, και είναι σημαντικός αυτός ο διάλογος, αλλά φαντάζομαι ότι ο κύριε Βάιντερ θα πει κάποια παρόμοια πράγματα. Κύριε Βάιντερε, ναι, σας ευχαριστώ. Εγώ ήθελα να ευχαριστήσω τον πρεσβευτή του Μπαχρέιν και να ευχαριστήσω και τους ε, συναδελφούς, τους βουλευτές του Μπαχρέιν. Διασφάλισαν ότι η δουλειά της αντιπροσωπείας θα εξελισσόταν ομαλά και νομίζω ότι κερδίσαμε φίλους και νομίζω ότι θα υπάρξει τώρα ένας ε, γνήσιος, ένας αυθεντικός διάλογος ε, και ότι θα υπάρχει ενοποίηση του λέω στον Παχρέν χωρίς συγκρούσεις. Ε, ήθελα να πω ότι ο κύριος στόχος μας ήταν να παρατηρήσουμε, να δώσουμε συμβουλές και να βοηθήσουμε. αυτό το ψήφισμα κατά κάποιο τρόπο δεν ήταν ισορροπημένο κατά την άποψή μου. Και νομίζω ότι η έκθεση αυτή είναι ισορροπημένη. Βασίζεται σε γεγονότα και πρέπει να εργαστούμε περαιτέρω υπό αυτή τη σκοπιά. Επίσης, ε, θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον κύριο Αμπτούλη Ραχμαν Ραχσίτ Μπουρτζάη ο οποίος ε, ήταν επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, πάντοτε συνόδευε την αντιπροσωπεία από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ και διασφάλισε στο να υλοποιηθεί ομαλά η δουλειά μας. Ο κύριος σε πολύ καλύτερα αγγλικά από τα δικά μου, εξέφρασε όσα ήθελα να πω για το ρόλο του Μπαχρέιν στην ευρύτερη περιοχή. Αν συγκρίνουμε τον Μπαχρέιν με άλλες χώρες ε, στην περιοχή, θα έλεγα ότι έχουμε πάρα πολύ καλές αφετηρίες και πρέπει να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας. Okay, now before I give the floor to Mr. just let... Λοιπόν, πριν να δώσω το λόγο στον Τόκης να σας πω ότι ευχαριστώ κύριε Πρεσβευτά και εσάς και την ομάδα σας για τις προετοιμασίες. Ευχαριστώ σας, σας το δώσω και γραπτός, μαζί με την έκθεση της αντιπροσωπίας. Κύριε Τόκης, σας παρακαλώ να είστε σύντομος γιατί έχουμε ξεπεράσει το χρόνο. Είμαι πολύ σύντομος. Πιστεύω ότι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η έκθεση της αντιπροσωπείας δεν έλαβαν χώρα την κατάλληλη χρονική στιγμή. Γιατί αν καταδικάζουμε τον Μπαχρέιν σε ένα ψήφισμα, τότε αποδυναμώνουμε την ενδιάμεση δουλειά της αντιπροσωπείας. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι είναι κρίμα που η έκθεση και το ψήφισμα έλαβαν χώρα ταυτόχρονα μήπως και επίσκεψη της προσωπίας, πρέπει να υποστηρίξουμε τον Μπαχρέιν να πετύχει τους στόχους του και να συνεργαστούμε καλύτερα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους για αυτή την αποστολή. Σας ευχαριστούμε για αυτή την πληρή έκθεση. Να περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα. Κύριε Βάγκαρε, με τη σας έχουμε τις επιπτώσεις και οικονομικής κρίσης στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η γραμματεία έχει λάβει 124 τροπολογίες. Από ό,τι καταλαβαίνω εργάζεστε επί συμβιβαστικών τροπολογιών. Και την επόμενη εβδομάδα θα συναντηθείτε και με τους κοιότητες εισηγητές. Κύριε εισηγητές είναι κύριε Βερσιά, κύριο Στάνοκο, κύριο Σταβάρες, κύριο Σάκε και κύριο Σμάρτη. Να ξεκινήσουμε δίνοντα το λόγο στην κυρία Βάιντερε και κατόπιν ε, θα ακούσουμε τους κοιοδησίτες. Παρακαλώ, εισηγήτρια. Αυτή τη φορά θα μιλήσω στη δική μου γλώσσα. Γιατί είναι δύσκολο να μιλάω τόσο πολλά αγγλικά. Θα μιλήσω λετωνικά λοιπόν. Ξέρετε, συνάδελφοι. Μόλις έφτασαν οι τροπολογίες των συναδέλφων στο email μου 124 τροπολογίες. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να ξεκινήσουμε, να συνεργαζόμαστε για να βελτιώσουμε την εκθέση αυτή. Και ολόψυχα, ελπίζω, Μάλλον ολόψυχα θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που έστειλαν τις τροπολογίες. Τις έχω εξετάσει και είμαι σίγουρη ότι περισσότερες πραγματικά θα βελτιώσουν την έκθεσή μου σε σχέση με την αρχική της μορφή. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν όλους τους συναδέλφους. Ίσως θα είχε νόημα να φερθούμε επί συγκεκριμένων τροπολογιών. Συζητήσαμε την εκθέση συνολικά σε περασμένη συνεδρίαση. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δουλειά σου. Ευχαριστώ και τους υπόλοιπους συναδέλφους που έστειλαν τις τροπολογίες. Βέβαια, δεν μπόρεσα να... Δεν θα μπορέσω τώρα να αναφερθώ και στις 124. Αλλά να πω ότι συμφωνώ με όσους ε, είπαν ε, ότι η διαφθορά έχει αρνητικό αντίκτυπο στο σεβασμό των ανθρωπινών δικαιωμάτων και εκπώνησα μία πρόταση συμβαστικής τροπολογίας. Ε, την ε, επόμενη εβδομάδα θα συναντηθούμε με όλους τους κοινούς συζητητές για να συζητήσουμε αυτές τις συμβιβαστικές τροπολογίες και θα δω ποια είναι τα επιχειρήματα πίσω από τις τροπολογίες. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, δεν βλέπω την κυρία Βερζιά εδώ. Χαίρομαι όμως βέβαια που είναι άλλοι συνάδελφοι, όπως ο κύριος Σταβάρες, κύριος Όμπιο. Όμως, ε, συμφωνώ με συναδέλφους που τόνισαν τον αρνητικό αντίκτυπο της διαφθοράς. Θέλω να αναφερθώ και στην Αναγκόμεση και στον κύριο Μάρτιν που κατέθεσαν κάποιες τροπολογίε προ αυτήν την κατεύθυνση. Ο κύριο Ταβάρες επίσης αναφέρεται στη διαφθορά. Θα προσπαθήσω λοιπόν να προσθέσω μια συμβαστική τροπολογία για το θέμα αυτό. Κάθε τροπολογία έχει το η λογική της. Εγώ θα προσπαθήσω να την αντικατοπτρίσω. Κατά τη διάρκεια της κρίσης είναι σημαντικό να τονίζουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αναπτυξική βοήθεια, όπως ε, τονίζεται στην τροπολογία 23. Και επίσης είναι σημαντικό να τονίσουμε πώς το κάνουμε αυτό. Ευχαριστώ κύριο ο οποίος ε, στην τροπολογία 74 το αναφέρει αυτό. Εγώ προσπάθησα αυτή την ιδέα να τη συμπεριλάβω και στη δική μου έκθεση. Στην τροπολογία 32, ο κύριο Ταβάρε ε, υπογραμμίζει ότι πρέπει να υποστηρίξουμε τι πολιτικές εξελίξεις στις τρίτες χώρες. Ακόμη και αν είναι δύσκολες οι οικονομικές συνθήκες. Και επίση κάποιο άλλο συνάδελφο ε, στην τροπολογία 71 τονίζει αυτό και συμφωνώ. Κυρία Γέγκλε, ήταν πολύ δημιουργική στην προσέγγιση της. Επίσης, με ανησυχούν τα προβλήματα που έχουν ε, οι κάτοικοι όταν ε, κάποιες μεγάλες εταιρείες ε, θέλουν να αγοράσουν τη γη τους. Ε, σας ευχαριστώ λοιπόν για τις τροπολογίες 49, 96 και 97. Θεωρώ και εγώ ότι η ανάπτυξη της γεωργίας και υποστήριξη της τοπικής παραγωγής είναι ένα σημαντικό στοιχείο σε κάθε στρατηγική. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στην τροπολογία 56. Συμφωνώ, το Ζαρουάτ. Πρέπει να βελτιώσουμε τον ανταγωνισμό των τρίτων χωρών. Αυτό τονίζεται στην τροπολογία 109. Ευχαριστώ και την κυρία Βερζιά, τον κύριο Όμπιο για τις τροπολογίες τους που τονίζουν πως ε, πρέπει να έχουμε μία επικοδομητική προσέγγιση και απέναντι στο δικαστικό σύστημα. Δεν θα μπορέσω να υποστηρίξω όλες τις τροπολογίες. γιατί κάποιες αναφερθήκαν σε στην κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ έχω πει ότι τα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που δεν έχουν να κάνουν με τα προβλήματα των χωρών δεν θα προσεγγιστούν εδώ. γιατί η κρίση έχει αγγίξει κάθε χώρα με διαφορετικό τρόπο. Έτσι λοιπόν ίσως ε, τα προβλήματα των κρατών μελών θα μπορούσαμε να τα αναλύσουμε σε άλλη έκθεση. Αν ε, ήταν εδώ η κυρία Βερζιά, θα της έλεγα ότι παρουσίασε πάρα πολλές τροπολογίες. Εγώ μπορώ να υποστηρίξω μόνο τις μισές από αυτές αλλά όχι τις, τις υπόλοιπες γιατί έχουμε και πολιτικές διαφορές. Έτσι λοιπόν μάλλον θα έχουμε τμηματικές ψηφοφορίες στην περίπτωση αυτή. Αν κάποιοι συνάδελφοι που βρίσκονται εδώ θα ήθελαν ε, να πούν δύο λόγια να σας πω ότι δεν μπορώ να τοποθετηθώ για τις ε, παραγράφους που προτείνονται προς διαγραφή. Θα ήθελα να ακούσω γιατί προτείνεται διαγραφή για κάποιες παραγράφους, γιατί δεν μπορούσα να καταλάβω σε ορισμένες περιπτώσεις. Αν κάποιοι από τους συναδέλφους που πρότειναν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες βρίσκονται εδώ, ίσως ε, θα μπορούσατε να μου δώσετε κάποιες εξηγήσεις. Ίσως ε, οι σκιώδεις εισηγητές να μπορούσαν να να μου αναλύσουν την αιτία του έτσι ώστε να μπορέσω να αποφασίσω. Όπως σας είπα, σας ευχαριστώ για τις 124 αυτές τις τροπολογίες. Αν αμφισβήτητα θα βελτιώσουν την έκθεση και θα έχουμε μια κοινή θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Παϊτήρη. Ήλεγξα Εάν μπορεί να έρθει η κυρία Βριζιά, αλλά δυστυχώ δεν μπορεί. Πάντω σίγουρα την επόμενη εβδομάδα στην προγραμματισμένη σα συνάντηση θα είναι και ο κύριο Οπιόλτ. αντικαθιστά τον κύριο Μάρτιν. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο, Πρόεδρε. Εδώ αντικαθιστώ τον Ντέβιντ Μάρτιν που είναι στην Ιορδανία σε αποστολή και είναι σκιώδης για την ομάδα μας. Έχουμε εκλογές στη χώρα εκείνη για το κατοκοινοβούλιο. Αυτή τη στιγμή νομίζω υλοποιούνται και μου ζήτησε να σας ζητήσω συγγνώμη για την απουσία του. Επίσης, ε, έρθει επαφή με κάποιον άλλο συνάδελφο για να παρουσιάσω εγώ τα σχολιά του. Μου είπε ότι γενικά κρίνει θετικά το κείμενο ότι μπορεί να αποτελέσει τη βάση ευρεία συνένεση. Κατά δεύτερον, δεν ε, βλέπει προβλήματα σε παραπάνω από 11 τροπολογίες που παρουσιάστηκαν. Ε, καθώς πρόκειται για εκθέσει πρωτοβουλία όμως θεωρεί ότι παρουσιάστηκαν πολλές ε, τροπολογίες. Τρίτον, αναμένει ότι σε μία συνεδρίαση με την εισηγήτρια να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε τροπολογία συμβασμού που να επιτρέψουν την ευρεία συνένεση και ότι είναι στη διάθεση της εισηγήτριας προς αυτή την κατεύθυνση. Ήταν πάρα πολύ εύκολο να κάνω αυτή τη σύνοψη γιατί συνάδει απόλυτα και με την προσωπική μου άποψη για την έκθεση. Σας ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε. Κύριο Σταβάρη, έχετε το λόγο. Με συγχωρείτε. Γιατί είχα ξεκινήσει να διαβάζω ότι ένας από τους ε, συγγραφείς της ε, διαβόητης μάλλον έκθεσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου μόλις απολύθηκε Βλέπετε λοιπόν με τι ποιότητα συντάσσονται οι εκθέσει του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου για ορισμένε από τι χώρε που περνάνε κρίση. Μπράβο, περιπτώσει. Ήταν ένα σχόλιο, α πούμε, ε, σχετικό γιατί όπως βλέπετε η κρίση δεν καθιστά μόνο ορισμένε, χώρες ευάλωτε αλλά όλους μας σε θεσμικό επίπεδο. Ε, ε, ε, ελπίζω ότι αυτή η έκθεση είναι πολύ καλύτερη από την άλλη του Δούνου του στην οποία αναφέρθηκα. Θεωρώ ότι αυτή η έκθεση έχει πολλές έξυπνες και σωστές προτάσεις. Έχω συνεισφέρει ορισμένες τροπολογίες, όχι πολλές γιατί θεωρώ προς ότι η έκθεση βρίσκεται προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι περισσότερες τροπολογίες που πρότεινα είναι περισσότερο σε, για λεπτομέρειες ή για να ασφαλίσω ότι αναφερόμαστε ότι αναφερόμαστε σε ζητήματα περιβάλλοντος ή άλλα θέματα που θεωρώ σημαντικά. Θέλω να είναι σαφές στην έκθεση ότι η κριτική που ασκούμε αφορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι Προφανέ ότι αυτό η κυρία Βάιντερ ήθελε να το εκφράσει, αλλά ήθελε να είναι σαφέ και στο κείμενο. Τρεις ε, πτυχές λοιπόν προσπαθώ να ε, αντιμετωπίσω με τις τροπολογίες με. Πρώτον, η τροπολογία 11 αφορά ακριβώς αυτό το ζήτημα. Αυτό που προσπαθώ να κάνω με την τροπολογία 11 λοιπόν είναι να πω ότι η κρίση μας έχει καταστήσει όλους πιο ευάλωτους, έχει καταστήσει την Ευρώπη περισσότερο ευάλωτη από οικονομική πλευρά, αλλά αυτό έχει επιπτώσει και στην εξωτερική πολιτική και στην πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κάτι που το βλέπω καθημερινά και στη χώρα μου την Πορτογαλία. Όταν μια κυβέρνηση ψάχνει απεγνωσμένα χρήματα, αναγκάζεται να εκποιήσει τη δημόσια περιουσία, πιθανώς ε, δημόσιες επιχειρήσεις σε χώρες οι οποίες να ε, ε, επισδικούνται από αυταρχικά καθεστώτα και δεν έχει την πολυτέλεια μια χώρα η οποία αναζητά έτσι ε, χρήματα να θέσει το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όταν προσπαθεί να κάνει ιδιωτικοποίησεις για παράδειγμα. Άρα η οικονομική κρίση βλέπετε πως έχει άμεσο αντίκτυπο στην εξωτερική μας πολιτική και στις πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ακολουθούμε. Δεύτερη τροπολογία που θέλω να, στην οποία θέλω να αναφερθώ, η 18, η σχέση μεταξύ της διαφθοράς και της διάβρωσης των δημοκρατικών θεσμών. Δηλαδή η υποχώρηση της πίστης των πολιτών στην νομιμότητα και στους δημοκρατικούς θεσμούς. Είναι επίσης ένα φαινόμενο που έχει ενταθεί εξαιτίας και μετά την οικονομική κρίση, μετά το 2008. Και θεωρώ ότι πρέπει να το αναφέρουμε. Από ό,τι φαίνεται όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Τρίτη τροπολογία, η 32, στην οποία αναφέρθηκε και η κυρία Βάιντερε. Τα άμεσα αποτελέσματα της κρίσης και η κρίση αυτή μπορεί να αναγκάσει τις κυβερνήσεις να περιορίσουν την ανθρωπιστική βοήθεια και την βοήθεια αναπτυξιακής συνεργασίας που παρέχουν. Κάτι που θα έχει δυσμενές αντίκτυπος τους στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας. Ήδη ορισμένες κυβερνήσεις στην Ευρώπη έχουν προχωρήσει σε οριζόντιες περικοπές πράγμα που έχει αγγίξει και την αναπτυξιακή βοήθεια. Αυτά είναι, αυτές είναι οι τρεις σημαντικότερες τροπολογίες που προτείνω και φυσικά βρίσκομαι στην διάθεση ε, της κυρίας Βάιντερε για να βρούμε ε, συμβιβαστικές λύσεις και συμβαστικές διατυπώσεις. Καθώς επίσης και με τις, στις συναντήσεις που θα έχουμε τις επόμενες εβδομάδες. Θα ήθελα να πω ότι αυτές οι τρεις τροπολογίες σε γενικές γραμμές πηγαίνουν στην ίδια κατεύθυνση με την τροπολογία 61 στα εκτιμώντας και είναι και ένα ζήτημα που είχε συζητηθεί και κατά την συζήτηση της δικής μου γνωμοδότησης και είναι το εξή ότι αν αρχίσουμε να κάνουμε εκπτώσεις στην εξωτερική μας πολιτική και την πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τι θα τις θεωρήσουμε ε, ρεαλιστικές, γιατί θα πούμε ότι πρέπει να, ε, ε, βραχυπρόθεσμα να είναι χρήσιμες. Αυτός ο εντός εισαγωγικών πραγματισμός στην πραγματικότητα μακροπρόθεσμα θα υπονομεύσει την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που επιδιώκουμε. Φαίνεται σαν τα ανθρώπινα δικαιώματα να είναι διακοσμητικά ξεχνούμε τις ίδιες τις συνθήκες που θέτουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ίδια τη βάση του οικοδομήματος, τη θεωρούν έναν από τους πυλώνες του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, όχι κάτι που απλώς προσθέτουμε στο τέλος διακοσμητικά. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης δεν θα πρέπει να κάνει εκπτώσεις παραχωρήσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί μακροπρόθεσμα αυτό θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα στι τρίτε χώρε, στα θύματα των παραβιάσεων ανθρώπινων δικαιωμάτων στι τρίτε χώρε, αλλά ε, αργότερα αυτό θα έχει ε, δυσμενεί επιπτώσει και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα υπονομευθούν τα πρότυπα, ε, τα κοινωνικά, τα πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα πρότυπα για το περιβάλλον. Και τελικά όλε οι αρχέ που θα θέλαμε να προστατεύσουμε για του Ευρωπαίου πολίτε, καταναλωτέ κτλ. πιστεύω ότι δεν περισσεύει ποτέ μια επανάληψη ακόμα αυτών των αρχών. Πρέπει να συνεχίσουμε να τα επαναλαμβάνουμε αυτά τα πράγματα προκειμένου να εφαρμοστούν τελικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ταβάρες. Ο κύριο Τάνοκ δεν είναι πια εδώ. Εξ όσων γνωρίζω δεν έχει προτείνει τροπολογίε. Την κυρία Σάρκε δεν με έχει ενημερώσει, αλλά είμαι βέβαιη ότι θα παραστεί στην συνάντηση τη επόμενη εβδομάδα των σκιώδων συγγητών. Θεωρώ επίσης ότι οι γνωμοδότηση που λάβατε από τον κύριο Τέιλορ θα ληφθεί υπόψη τι τροπολογίε που εκείνος θα προτείνει. Εάν υπάρξουν σοβαρά προβλήματα θα ήθελα να το γνωρίζω γιατί ήδη έχουμε ξεκινήσει σημαντικές συζητήσεις με τον κύριο Τέιλορ για μια άλλη έκθεση και επιθυμούσα, αν είναι δυνατόν, να ενσωματωθούν όλες τις τροπολογίες του Ντέιβιτ σε αυτήν την έκθεση. Ο κύριος Φαν έχει ζητήσει τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς τώρα μελετάμε τις τροπολογίες, δεν θα ασπεύσω να σχολιάσω. Ελπίζω να μην πειράζει αλλά θα ήθελα να πω κάτι που θα το θέσουν και οι μη κυβερνητικέ ή θα το έθεταν αν ε, μπορούσαν να μιλήσουν. Μια πρωτοβουλία που αρχίσαμε μόλις σήμερα το πρωί και που μπορεί να ενδιαφέρει την εκθεσή σας. Πρόκειται για το, την εκστρατεία αρκετά τρόφιμα αν. 100 μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, σε σχέση με την συνάντηση των G8 αργότερα μέσα σε αυτό το χρόνο. Θα ήθελα να το αναφέρω αυτό γιατί αποτελεί μια μεγάλη πρωτοβουλία. Ευχαριστώ κυρία Σουάνη. Κυρία Βαϊντέρ θα κλείσει τη συζήτηση. Θέλω να πω ότι είμαι ευγνώμων για τις τροπολογίες σας που είναι πολύτιμες και ε, τα σχόλιά σας επίσης και περιμένω την επόμενη εβδομάδα τώρα για να οριστικοποιήσουμε τη δουλειά μας με τις συμβιβαστικές τροπολογίες. και ελπίζω να είναι και στο μέλλον τόσο επικοδομητική η δουλειά όσο ήταν μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Τώρα, από εδώ και πέρα τι θα γίνει. Την επόμενη εβδομάδα η μετά θα εξετάσουμε τις τροπολογίες στην ΑΦΕΤ στις 18 Φεβρουαρίου. Η ψηφοφορία θα είναι 19 Φεβρουαρίου στην ΑΦΕΤ και θα πάει στην Ολομέλεια του Απριλίου όπου θα εγκριθεί η έκθεση. Ευχαριστώ. Και τώρα περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι η έκθεση της αντιπροσωπείας δρούα στην Τουρκία. Η, α, η κυρία Περζιά θα έρθει. Θα έρθει. Η κυρία Βαρζιά και εγώ είμαστε τα μέλη της αντιπροσωπείας για την Τουρκία που είχε διπλό νόημα και αποστολή γιατί πήγαμε μια μέρα στην Άγκυρα και είδαμε διάφορα υπουργεία και τη οργανώσεις της ε, κοινωνίας των πολιτών και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και μετά πήγαμε στα τουρκο-συριακά σύνορα. Επίσης έχετε πρόσφατα τη γραπτή μας έκθεση, μόλις ε, ε, έχει διανεμηθεί, είναι φρέσκια φρέσκια. Ε, στην αρχή της συνεδρίασης την διανύμαμε και τώρα προτιμώ να περάσω στα γερμανικά διότι θα χρησιμοποιήσω τις σημειώσεις που κράτησα. Τα κεντρικά θέματα για μας κατά την αποστολή ήταν η κατάσταση με την ελευθερία μέσων ενημέρωσης και ελευθερία μέσων, ε, μεταρρυθμίσεις στη δικαστική εξουσία, δηλαδή τα διεθνή πρότυπα πώς μεταφέρονται στο εθνικό δίκαιο, η πολιτική πώς επηρεάζει την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, Μόλις φτάσαμε συναντήσαμε εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών από 13 διαφορετικές οργανώσεις ε, στην αρχή και διαρκώς ακούγαμε ανεξάρτητα αν ήταν συνδικαλιστές, αν ήταν γυναικείες οργανώσεις, αν ήταν δημοσιογράφοι, αν ήταν οργανώσεις ΛΟΑΔ, λεσβείες ομοφιλόφιλοι κλπ. Όλοι μας λέγανε ότι στην Τουρκία Γίνεται πολλή δουλειά σε, σε επίσημο επίπεδο για την εναρμόνιση νομοθεσίας ή τη βελτίωση των θεσμών. Για παράδειγμα, στον τομέα των δικαιωμάτων των γυναικών αναγνωρίζεται ότι δεν έχουμε αρκετά τηλέφωνα κλήσεις ε, που μπορούν να χρησιμοποιούν γυναίκες με προβλήματα ή στέγη που θα προστατεύει τις κακοποιημένες γυναίκες. Αυτό είναι θετικό λοιπόν ότι το κοιτάζουν. Παράλληλα βλέπουμε όμως ότι η πολιτική ηγεσία δεν βλέπει με πολύ καλό μάτι ότι γίνονται πράγματα εκτός ελέγχου της ε, στα, στα δικαιώματα των γυναικών. Είναι λυπηρό για παράδειγμα, πολύ λυπηρό, ότι διαγράφησαν κάποιοι τίτλοι γυναικών από το Υπουργείο που είναι υπεύθυνο για την προστασία της οικογένειας και της κοινωνικής ευημερίας και αυτό ε, δείχνει, και το είδαν οι οργανώσεις, μια διαφορετική σκέψη ότι τα δικαιώματα δικαιών τα βλέπουν πάντοτε στα πλαίσια του μορφώματος της ε, παραδοσιακής οικογένειας. Ένα άλλο θετικό βήμα είναι ότι υπάρχουν ε, τώρα καινούργιες ε, οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και έχουν οριστεί τα μέλη της οργάνωσης και θα πρέπει να ε, δημιουργήσουν, να συγκροτήσουν ένα σώμα με πρόεδρο κλπ. Δεν ξέρουν όμως πότε ακριβώς θα γίνει αυτό. Η κριτική που γίνεται σε αυτό το θεσμικό όργανο για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, αφορά την εντολή τους και τον τρόπο εργασία τους, εργασίας τους που δεν ανταποκρίνεται στο, στις προδιαγραφές των ε, Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την ανεξαρτησία τους θα πρέπει να δούμε όλα τα θεσμικά όργανα που ε, αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχουν ε, έρευνες και μελέτες σχετικά με τα, τα ιδρύματα αυτά και τους θεσμούς που υπάρχουν στην Ανατολική Ευρώπη. Παντού πρέπει να τα δούμε για να δούμε αν είναι ανεξάρτητα. Εμείς ε, μιλήσαμε και με κυβερνητικούς εκπροσώπους στην Τουρκία και μας είπαν ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι όλα τα ε, όργανα ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεσμοί, δεν είναι όλα στο ίδιο επίπεδο. Έτσι λοιπόν ε, πρέπει να με το έργο του Ινστιτούτου αυτού στην Τουρκία. Δύο εβδομάδες μετά την έναρξη των εργασιών, ο διαμεσολαβητή ο διαμεσολαβητής άρχισε επίσης να λειτουργεί. Ε, ασχολείται με προσφυγές και καταγγελίες που του υποβάλλουν Τούρκοι πολίτες, είτε πρόκειται για λάθη, για αυθαιρεσίες στη διοίκηση και στις αρχές. Είναι λοιπόν μια πολύ σημαντική υπηρεσία που προασπίζει ανθρώπινα δικαιώματα, ε, θεμελιώδη δικαιώματα, καταπολεμεί τη διαφθορά και νομίζω ότι ένα μεγάλο πρόβλημα ε, αφορά το διορισμό του ίδιου του διαμεσολαβητή. Γιατί αποφάσισαν ότι ο προηγούμενος, ο, ο πρώην δικαστής ε, κ. Σιμερόγλου θα αναλάμβανε τη θέση αυτή. Μιλήσαμε μαζί του, αλλά στην ανάληψη του δημόσιου αξιώματος και ε, στην κριτική που γίνεται αναφέρεται ότι συμμετείχε στο ακυρωτικό δικαστήριο σε ε, μια δίκη που έβγαλε απόφαση κατά του Χραντ Ντίνκ, ενός ε, Αρμένιου δημοσιογράφου και είναι τραγικό και ατυχέστατο το γεγονός ότι ο Χραντ Ντίνκ αργότερα δολοφονήθηκε. Και αυτό στις συνομιλίες μας οδήγησε σε πολλές επιφυλάξεις. Αν δηλαδή ε, οι τουρκικές αρχές βλέπουν ε, με θετικό μάτι την ανεξαρτησία του διαμεσολαβητή. Ο κύριος Σιμερόγλου είπε ότι τελείως έμεσα είχε ασχοληθεί με την υπόθεση που σας ανέφερα. Αλλά βεβαίως δεν μπορούσε και να ισχυριστεί ότι δεν είχε καμία σχέση. Θα αναφέρω και κάτι ακόμα γιατί δύο μέρες πριν φτάσουμε στην Τουρκία ο Πρωθυπουργός Ερδογάν επίσημα σε μια ομιλία του είπε ότι θεωρεί ότι η διάκριση των εξουσιών δεν είναι ότι καλύτερο πάντα για την Τουρκία. και εκπρόσωποι των επιστημών και της κοινωνίας των πολιτών ε, σχολίασαν αυτήν την ε, αναφορά. Γιατί ε, αν αναφέρεται ένας Πρωθυπουργό σε τέτοια θεμελιώδη ζητήματα και τα αμφισβητεί όπως τη διάκριση των ε, εξουσιών αυτό οδηγεί σε πολλές συζητήσεις και τα παραδείγματα που συζητήσαμε σε σχέση με την άσκηση επιρροής στη δικαστική εξουσία ε, το δείχνει αυτό καθαρά. Έχουμε την υπόθεση Πίνα Σέλικ που είναι μια κοινωνιολόγος, φεμινίστρια και συγγραφέας που κατηγορήθηκε το 1998 ότι συμμετείχε στην ε, Κωνσταντινούπολη σε μια βομβιστική επίθεση. Ακολούθησε μια μακρά δικαστική διαδικασία, συνελήφθη, βασανίστηκε ε, στη φυλακή. Τρεις φορές αθωώθηκε εντωμεταξύ από διαφορετικά, τρία διαφορετικά δικαστήρια. Το φθινόπωρο όμως ένας δικαστής που συμμετείχε στην διαδικασία ασθένησε και αντικαταστάθηκε από καινούριο. Και τώρα επίκειται κατά δίκη ίσως και για διαβίου φυλάκιση ε, Σόβια. Την περασμένη εβδομάδα ε, συζητήθηκε το θέμα στην αντιπροσωπεία ε, με την Τουρκία. Αύριο αναμένεται η απόφαση. Και δεν... Τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει μία προσπάθεια πολιτικής παρέμβασης στη δικαστική εξουσία. Εδώ προστίθεται κάτι ακόμα που θα το αναφέρω παρόλο που το είδαμε στις 18 Ιανουαρίου ε, υπήρξε σειρά συλλήψεων δικηγόρων που είναι συνήγοροι ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πάντοτε όποτε υπάρχει αυτή η καταγγελία στο δικαστήριο Όποτε υπάρχουν κατηγορίες που αφορούν την ανεξαρτησία του λόγου, πάντα ασκούνται επιρροές ε, όταν αναφέρονται ε, τέτοια δικαιώματα. Ε, σε μια ενέργεια της αστυνομίας συνελήφθησαν για μιας 15 δικηγόρους. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο αυτό. Και έτσι στη δουλειά μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία θα πρέπει αυτά να τα παρακολουθούμε. Και ε, ε, βέβαια, ε, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης είδαμε ότι πραγματικά γίνεται μεγάλη προσπάθεια μεταφορά στην εθνική νομοθεσία διεθνών προτύπων και παρακολουθούνται και μεμονωμένες υποθέσεις και αποφάσεις από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ώστε να τα λαμβάνουν υπόψη στην εθνική νομοθεσία. Και γενικά παρακολουθούν το δικαστήριο γιατί... Οι περισσότερες υποθέσεις είναι από Τουρκία και Ρωσία. Όμως θα έλεγα ότι δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε τις πολιτικές παρεμβάσεις στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, της δικαστικής εξουσίας. Ένα άλλο θέμα αφορά τους Κούρδους, άνδρες και γυναίκες. Εδώ βεβαίως είναι σημαντική η ένοπλη αντιπαράθεση. Ε, είχαμε τις εκλογές το 2011, το 2012 δεν πέρασε μέρα σχεδόν ε, κατά το περσινό έτος χωρίς να λάβει χώρα μια βίαιη αντιπαράθεση. Ε, μένα ήταν η πρώτη μου επίσκεψη στην Τουρκία ως μέλος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και με εντυπωσίασε η κατάσταση εκεί, δικαίου. Όταν οποτεδήποτε συζητείται η κατάσταση των Κούρδων, ανεξάρτητα από το επίπεδο, στο Υπουργείο, το πλαίσιο, πάντα χρησιμοποιείται η λέξη τρομοκράτης ε, για να χαρακτηρίσει τους Κούρδους, άνδρες, γυναίκες, ακτιβιστές. Αυτό το πράγμα με έκανε να απορρίσω διότι, και με ξένησε, διότι ε, θα πρέπει να δούμε ποια, ε, ε, γιατί αντιμετωπίζονται, τι θέσεις ακριβώς παίρνουν οι Κούρδοι. Ε, υπάρχει διαφοροποίηση. στο Εθνικό Κοινοβούλιο αρνούνται να καταλάβουν τις θέσεις τους οι βουλευτές λόγω της σύλληψης έξι συναδέλφων. Εμείς κάναμε και συζητήσεις με βουλευτές του κόμματος 5 και είναι πολύ απεσιόδοξη σε σχέση με την τροποποίηση του συντάγματος εδώ, ε, ούτως ώστε να βελτιωθούν τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων. Και είναι δύσκολο να δούμε πώς μπορεί να αλλάξει το όριο του 10% που ισχύει για τις βουλευτικές εκλογές. Πρέπει λοιπόν να τύχει επεξεργασία του συντάγματος ε, και αυτό στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πρέπει να το παρακολουθούμε και να βλέπουμε αν υπάρχουν ε, ακροάσεις, ε, δηλαδή δίκες κατά συνηγόρων ακτιβιστών ή των ακτιβιστών των ίδιων και θα πρέπει να φροντίζομαι να δίνεται δημοσιότητα σε αυτές τις υποθέσεις. Συναντήσαμε και τον Υπουργό Υπεύθυνο για Ευρωπαϊκά Θέματα ο Υπουργός διαμαρτυρήθηκε έντονα γιατί δεν βλέπει ε, πρόοδο από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υπάρξει ενεργός ε, ατζέντα ε, προσχώρησης. Είπε ότι ελπίζει να εντατικοποιηθούν οι διαδικασίες επί Ιρλανδικής Προεδρίας και να ανοίξει τουλάχιστον ένα ακόμη κεφάλαιο. Ένα θέμα που θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε και με την αντιπροσωπεία με την Τουρκία είναι να δούμε μήπως μπορούν να ανοίξουν τα κεφάλαια 23 και 24 που αφορούν την τουρκική δικαιοσύνη και την ε, προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μήπως υπάρξει κάποια κινητικότητα εκεί. Εμείς ε, θα ασχοληθούμε τότε εντατικά με αυτά τα θέματα στην ε, Επιτροπή μας. Είχαμε συναντήσει και στο Κοινοβούλιο με την Επιτροπή για την Εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση αυτή και δεν είμαστε μόνο εμείς οι δύο εκεί. Μέσω ημών ε, προσεκλήθησαν και όλα τα μέλη της Επιτροπής να συμμετάχουν σε πολλές εκδηλώσεις στην Τουρκία και σε πολλές ε, πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί θα γίνει μια σειρά διασκέψεων μεταξύ Ευρωπαίων και Κούρδων βουλευτών και μπορούν να είναι και εθνικοί βουλευτές για την ε, ορθή διακυβέρνηση, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και τέτοια θέματα. Αυτά λοιπόν σε σχέση με τις συναντήσεις ε, που είχαμε στην Άγκυρα. Πρέπει να πω ότι η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Άγκυρα μας βοήθησε πάρα πολύ. Ιδιαίτερα το Human Rights Focal Point στην Άγκυρα που ήταν σημαντικό για την επιτυχία με τις συναντήσεις που είχαμε με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και με τα διάφορα Υπουργεία και το Κοινοβούλιο. Ε, είχαμε και ένα πρακτικό πρόβλημα οργανωτικό εκεί, γιατί θέλαμε να πάμε στα τουρκοσυριακά σύνορα. Δεν το επέτρεψε όμως η ομίχλη αυτό. Έπρεπε λοιπόν να αλλάξουμε το πρόγραμμα και πήγαμε στα Άδανα με το αεροπλάνο και μετά με το οδικός το βράδυ πήγαμε ακολουθήσαμε το άλλο μας το πρόγραμμα και ευχαριστούμε πολύ και την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, η κατάσταση στα τουρκο-συριακά ε, σύνορα ήταν πολύ εντυπωσιακό που είδαμε ότι περίπου 200.000 έγιναν δεκτοί σε καταβλισμούς ως πρόσφυγες από την τουρκική κυβέρνηση. Απλή καταβλισμοί, αλλά καλά εξοπλισμένοι για να καλύπτονται οι βασικές ανθρώπινες ανάγκες. Ο καταβλισμός που επισκεφθήκαμε έχει πολύ καλή υποδομή. Δηλαδή προπτικά έχει τη δυνατότητα αυτό διαχείρισης από τους πρόσφυγες που συμμετέχουν στην ε, ζωή του καταβλισμού. Υπάρχουν σχολεία, υπάρχουν υπηαγωγεία, υπάρχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Πολύ εντυπωσιακά όλα αυτά. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω και με τον διοικητή του Γκαζιαντέπ, εκεί πήγαμε, μέσω Άδανα, και είδα ότι ε, προσεγγίζουν καλά τα θέματα αυτά. προβλέπουν ότι δεν θα γυρίσουν οι πρόσφυγες σύντομα στην πατρίδα τους και η Τουρκία ε, προσαρμόζεται για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα να τους φιλοξενήσει. Υπάρχουν και πρόσφυγες που φιλοξενούνται από οικογένειες και δεν έχουν ε, επισήμως καταχωριστεί. Ε, η Τουρκία τώρα επεξεργάζεται ε, ειδικό νόμο περί ασύλου, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, αλλά αν κάποιος δεν είναι καταχωρισμένος, δεν δικαιούται κοινωνική βοήθεια, πράγμα που δυσκολεύει πολύ την κατάσταση μακροπρόθεσμα. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά όργανα της μπορούν να παράσχουν ανθρωπιστική βοήθεια, πρέπει να βρουν έναν τρόπο να βοηθήσουν αυτή την κατηγορία προσφύγων είτε μέσω διεθνών είτε μέσω εθνικών μη κυβερνητικών οργανώσεων εκεί. Πάρα πολύ δύσκολη είναι η κατάσταση των προσφύγων που ακόμα δεν μπόρεσαν να περάσουν τα ε, στην Τουρκία από τα τουρκοσυριακά σύνορα. Ε, πολλές φορές, ε, εμείς πήγαμε τέλος Δεκεμβρίου εκεί και μάθαμε ότι υπάρχουν σκηνές χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. απευθυνθήκαμε στην Επίτροπο Γεωργίευα, μάλλον θα αποστείλουμε επιστολή στην ε, Επίτροπο για να προσπαθήσει να ξεπεράσει και να λύσει τα γραφειοκρατικά προβλήματα που υπάρχουν, ούτω ώστε απευθείας να υποστηριχθεί η τουρκική κυβέρνηση ή μια μη κυβερνητική οργάνωση που στηρίζει τους πρόσφυγες με τρόπο καθόλου γραφειοκρατικό ή ελάχιστα γραφειοκρατικό και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τους υπόλοιπους πρόσφυγες που δεν τους έχουμε ακόμα καλύψει. Στο ίδιο το, στον ίδιο τον καταβλισμό κάναμε συζητήσεις με Σύριους ε, πρόσφυγες και μετά κάναμε, έκανα συζήτηση και με μια Συριακή Οργάνωση Νεολαίας. Το θέμα δεν ήταν τόσο πώς ζουν εκεί στον καταβλισμό, αλλά ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να μην παρέμβουν με τρόπο τέτοιο στη σύγκρουση ώστε ε, να ε, ε, συνεχίσει η κυβέρνηση να βομβαρδίζει τον ίδιο της τον πληθυσμό, τον ίδιο το λαό. είπα ότι μπορεί η στρατιωτική επέμβαση να κλιμακώσει την ένταση. Όλοι οι συνομιλητές είπαν ότι αυτό ε, δεν τους βρίσκει σύμφωνος. Νομίζουν ότι αυτό είναι μία ε, αυταπάτη. Ήταν καλό που έκανε την επίσκεψη αυτή η αντιπροσωπεία της Επιτροπής των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Λυπάμαι διότι στην διάσκεψη όλων των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών στις αρχές Δεκεμβρίου δεν μπόρεσαν να υιοθετήσουν ένα ειδικό πρόγραμμα ε, φιλοξενίας σύρων προσφύγων γιατί δεν ξέρω ποια λέξη να χρησιμοποιήσω ε, είναι ε, πολιτική καλής γειτονίας ε, το γεγονός ότι η Τουρκία ε, υποδέχεται τόσους πρόσφυγες αλλά δεν θα μπορέσει να συνεχίσει γιατί υπάρχουν και πολλοί τραυματίες ε, πολέμου. Πρέπει λοιπόν να υπογραμμίσω και εγώ και να αναδείξω το αίτημα αυτό που υπάρχει ότι μέσα από ένα resettlement program η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει και να βοηθήσει και την Τουρκία και άλλες γειτονικές χώρες όπως την Ιορδανία ή τον Λίβανο ώστε να υποδέχονται τους πρόσφυγες διότι πρέπει να υπολογίζουμε ότι δεν θα τελειώσει η αντιπαράθεση αυτή γρήγορα και θα πρέπει χρόνια ίσως να παραμείνουν οι πρόσφυγες στις χώρες που τους φιλοξενούν. Αυτά λοιπόν, η κυρία Βερζιά δεν ήρθε, φαίνεται ότι δεν μπόρεσε για να συμπληρώσει, να έρθει να συμπληρώσει. Εγώ ε, έκανα αυτή την έκθεση στην ε, ε, αντιπροσωπεία για την Τουρκία. Επίσης στην ΑΦΕΤ θα υποβάλουμε τη γραπτή μας έκθεση και θα δούμε τι ενδεχομένως ποιες τροποποιήσεις θα πρέπει να γίνουν. Τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Ομπιόλς, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για την ενημέρωση σε σχέση με την επίσκεψη της αντιπροσωπείας και σας ευχαριστούμε και για το έγγραφο. Θα το διαβάσω πολύ προσεκτικά γιατί είμαι σκιώδης εισηγητής για την ομάδα μου σε σχέση με την ετήσια έκθεση αξιολόγηση τη διαπραγματευτική διαδικασία για την προσχώρηση της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να κάνω ένα σύντομο σχόλιο σε σχέση με το συγκεκριμένη προβληματική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία. Βασικά, συμφωνώ με τη δική σας ερμηνεία της κατάστασης, όπως ε, την είδατε εκεί. Βέβαια, το βασικό ζήτημα είναι <laughs> αν θα θεωρούμε το ποτήρι μισοάδιο μισογεμάτο. Και προς αυτή την κατεύθυνση μια προβληματική κατάσταση θα πρέπει να μας οδηγήσει στο να είμαστε προσεκτικοί για το αν η τάση βελτιώνεται ή επιδεινώνεται. Δηλαδή δεν μπορούμε μόνο να λαμβάνουμε μία φωτογραφία μιας κατάστασης που σε πολλές πτυχές παρουσιάζει προβλήματα. Όμως εγώ θέλω να αφαιρθώ στη δική μας στάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στην εσωτερική κατάσταση της Τουρκίας και της ε, τάσης προς εξέλιξη. Όσο και αν προσπαθούμε στο διάλογο, στον εντοπισμό προβλημάτων, στην καταγγελία κάποιων προβληματικών καταστάσεων, στο να διαμαρτυρόμαστε ενώπιον τέτοιων καταστάσεων, αν δεν έχουμε μία στάση ελαχίστως συνεπούς για τη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας πιθανότητα δεν θα είμαστε ιδιαίτερα αποτελεσματικοί και νομίζω ότι μπορεί να είμαστε και αντιπαραγωγικοί δηλαδή μπορεί να προκαλέσουμε κάποιες συνέπειες που δεν επιθυμούμε αν επιθυμείτε συνέπειε, αναφέρομαι στο εξή. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε το 2005 να ξεκινήσει μια διαπραγματευτική διαδικασία για την προσχώρηση της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κατόπιν η διαδικασία αυτή πρακτικά λοκαρίστηκε. Νομίζω ότι οποιαδήποτε συνεπή στάση για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και θα πρέπει να οθεί προς το να γίνει κάθε δυνατό για να διατηρούμε ένα κοινό πολιτικό κριτήριο που να συνίσταται στην τήρηση της κλασικής αρχής pacta sunt servante. Συμφωνίες πρέπει να τηρούνται. Δηλαδή ότι αν ξεκίνησε μια διαπραγματευτική διαδικασία πρέπει και να ολοκληρωθεί. Εγώ νομίζω ότι το 2013 αποτελεί μια ευκαιρία να απεμπλοκαριστεί η κατάσταση αυτή. Έχουμε αλλαγή στη Γαλλία που είναι σημαντική γιατί βλέπουμε μια μετακίνηση παραδείγματος ε, της ε, κυβερνητικής ε, θέσης για το θέμα της Τουρκίας από θέσεις που βασίζονταν σε κριτήρια ιστορικά, σε κριτήρια πολιτισμού, θρησκευτικά κριτήρια. Ο προκάτοχος ε, του κ. Λέντε μας ε, είπε πολλές φορές ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δημιουργηθεί ένα σύστημα αξιολόγησης με οικονομικούς και πολιτικούς όρους συγκεκριμένου. Και όχι να μπαίνουμε σε άλλου είδους συζητήσεις. Ο στόχος ε, θα είναι να απεμπλοκαριστούν διαπραγματεύσεις, κυρίως σε ένα θέμα που αδιαφέρει ιδίως αυτή την υποεπιτροπή και έχει να κάνει με την απεμπλοκή των διαπραγματεύσεων στα κεφάλαια 23 και 24. Μιλάμε για τα κεφάλαια δικαιοσύνη, ανθρώπινα δικαιώματα, ελευθερία και ασφάλεια. Εγώ νομίζω ότι οποιαδήποτε αξιολόγηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία δεν ε, μπορεί να μην λαμβάνει υπόψη ιστορικά αυτό το μπλοκάρισμα και τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το αίτημα προσχώρησης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ε, ξέρετε ότι εντάσσεται σε μία δραματική συγκυρία. Η πρόεδρος αναφέρθηκε σε αυτό ότι έχουμε χιλιάδες πρόσφυγες από τη σύραξη της Συρίας σε τουρκική επικράτεια. Αν δεν υπάρξει συγκεκριμένη δέσμευση και αλληλεγγύη από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ζήτημα αυτό, η δική μας δουλειά για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα θα είναι πράγματι πολύ δύσκολη. Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Μπιόλς. Να δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Βερζιά. Και μήπως θα θέλετε να μας ουσιαστείτε και τη δική μας σας ε, άποψη. Και αν μπορείτε να απαντήσετε και στον κύριο Μπιόλς που είπε, ποια τάση μπορούμε να δούμε Ποια τάση μπορούσαμε να δούμε σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτή τη διμερή επίσκεψη. Διάβασα την τελική έκθεση και σε μεγάλο βαθμό συμφωνώ, συγγνώμη. Δεν μπορούσα να ακούσω τόσο είπατε γιατί έφτασα καθυστερημένα. Ένα από του συνεργάτε μου γενικά μου συνόψισε τόσα είπατε. Θεωρώ ότι δεν αναφέρεται ευρέως στο κουρδικό. Και αυτό το ζήτημα αναφέρθηκε ευρέως από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις που συναντήσαμε επί εγώ ξέρετε τι, επειδή ξέρετε και τι συνέβη στο Παρίσι με την δολοφονία των τριών ε, Κούρδων γυναικών ε, ήταν 50 ετών περίπου, επομένως ε, ευαισθητοποιήθηκα πάρα πολύ για το θέμα αυτό. Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με τα όσα μόλις είπατε. από του κυβερνητικού συναντητέ μας, εγώ κατάλαβα ότι τελικά δεν κατανοούσαν πολύ καλά τη στάση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό σε μεγάλο βαθμό συμφωνώ με τα όσα είπατε. Γιατί η Ευρωπαϊκή Θεσμή και κυρίως το Συμβούλιο των Υπουργών έχει μια ιδιαίτερα ασυνεπή στάση απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Γιατί ενέκρινε την υποψηφιότητα της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα δεν ε, μεταχειριστεί την Τουρκία όπως μεταχειριστήκε τις υπόλοιπες υποψήφιες χώρες. Τα κεφάλαια 23 και 24 είναι ουσιαστικά, είναι ουσιαστικά και δική μας ε, υποεπιτροπή και νομίζω ότι ουσιαστικά αυτό που βαρύνει ε, είναι αυτό που βαρύνει περισσότερο για τη δυνατότητα προσχώρησης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα θέματα που αναφέρατε με κάλυψαν, γιατί η εικόνα που μας παρουσιάστηκε στην Τουρκία σχετικά με το πώς εξελίσσεται το κράτος δικαίου, δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, για να χρησιμοποιήσω την ευρωπαϊκή ορολογία, είναι δραματικού χαρακτήρα. Μας ανέφεραν ότι υπάρχουν 8-10 πολιτικοί κρατούμενοι στις τουρκικές φυλακές και εξελίσσεται η καταστολή. Η φυσική καταστολή, οι Κούρδοι εκλεγμένοι, και όχι μόνο. Υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα που πρέπει πραγματικά να συζητηθεί στα πλαίσια του θέματος της προσχώρησης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι τα πράγματα μπερδεύονται ακόμη περισσότερο. Αλλά αν μου επιτρέπετε, Πρόεδρε, θα ήθελα να προσθέσω δύο λόγια σε σχέση με τις ε, συνέπειες που προκαλούνται από τη δολοφονία των γυναικών στο Παρίσι, γιατί νομίζω ότι κατόπιν ε, της απεργίας πείνας ε, στις τουρκικές φυλακές έχει ξεκινήσει ένας διάλογος μεταξύ της κυβέρνησης της Τουρκίας και του κυρίου Τσαλάν και τα δραματικά γεγονότα της Γαλλίας δεν θα πρέπει να βαρύνουν αυτή την ειρηνευτική διαδικασία. Εγώ χαίρομαι που έχουμε στην ημερήσια διάταξη προγραμματίσει μια συζήτηση στην επόμενη Ολομέλεια στο Στρασβούργο, γιατί νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ασκήσει όλο του το βάρος, όπως το έχει κάνει σε ορισμένα θέματα, δεν το πράττει πάντα, αλλά σε ορισμένα θέματα το έχει πράξει, γιατί πραγματικά έχει νόημα για όλους όσους ζουν στην τουρκική επικράτεια, για όλες τις εθνοτικές μειονότητες, αλλά και για όλο τον τουρκικό πληθυσμό. και κατά τα λοιπά θεωρώ ότι συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με την εκθεσή σας που είναι αρκετά Σε Ένα σημείο σημαντικό είναι ότι περίμενα περισσότερη απόκληση μεταξύ των ε, δύο εκπροσώπων ε, της αντιπολίτευσης που συναντήσαμε, αλλά αυτό που με εξέπληξε ήταν η σύγκληση απόψεων που μας προσίασαν. σε σχέση με το πώς αξιολογούσαν τις δημοκρατικές εξελίξεις και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη συζήτηση για το Σύνταγμα. Εγώ νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό το θέμα και θα έπρεπε να το επισημάνουμε. Ευχαριστώ κύριε Βερζιά. Νομίζω ότι μπορούμε να μπλουτίσουμε την έκθεση και να αναφέρουμε τι συζητήσαμε για το κουρδικό. Επίσης ξέχασα να σας πω ότι πολύ συχνά ε, μιλάμε για μια τεράστια απεργία πείνας. Νομίζω ότι πάνω από 600 άνθρωποι συμμετείχαν στην απεργία πείνας, νομίζω κυρίως Κούρδοι κρατούμενοι. Και Νομίζω ότι ήταν κατόπιν παρατήρηση και του ίδιου του Τσαλάν, αλλά ακούσαμε ότι και ο Υπουργό Δικαιοσύνη συνέβαλε στο να βρεθεί μια καλή λύση για να τελειώσει η απεργία πείνα. Μόλι το συνόψισε αυτό και νομίζω ότι και στην έκθεση θα μπορούσαμε να το αναφέρουμε. Επίση, να αναφερθούμε και στι διάφορε απόψει ε, των ομάδων τη αντιπολίτευση. Και πριν να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο τη Κομισιόν, να πω δύο λόγια στον κύριο Μπιόλ. Άκουσα προσεκτικά τι είπατε. Ρωτήσατε ποια είναι η τάση. Μία τάση είναι κάτι παραπάνω από αυτό που μπορεί να μάθει κάποιο ε, σε μία-δύο ημέρε ε, συνεδριάσεων. Εγώ προσωπικά παρακολουθούσα τη συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία απ' έξω, διαβάζοντα κτλ. Και, και πραγματικά ανησυχούσα πάρα πολύ για το πόσο ανοιχτά η κοινωνία των πολιτών έλεγε ότι υπάρχει ένα κενό σε σχέση με το τι υπάρχει στα χαρτιά, στα νομικά χαρτιά και με μονομενή αύξηση επιθέσεων κατά μονομένων ανθρώπων, κατά δημοσιογράφων, κατά ιδρυμάτων που είναι φιλικά προς τους Κούρδους. Αυτό το χάσμα συνεχίζει να μεγαλώνει. Έτσι λοιπόν, ε, εγώ αισθανθήκα ότι θέλω να μάθω περισσότερα για τα θέματα αυτά και μία από τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών έκανε μία πρόταση να επικεντρωνόμαστε μερικές φορές, δηλαδή ίσως και εκτός σύνθεσης να έχουμε ένα συγκεκριμένο σεμινάριο στις Βρυξέλλες για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έτσι ώστε να ενημερωνόμαστε και όχι μόνο να περιγράφουμε τα περιστατικά, αλλά να βλέπουμε και ποιες είναι οι τάσεις. Και νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε πιο ενεργοί, να έχουμε ένα πιο ισχυρό διάλογο με το κοινοβούλιο στην Τουρκία, την κυβέρνηση, την κοινωνία των πολιτών. και θα ήθελα να αυξήσουμε τις προσπαθίες μας ε, για να ξεκινήσουν πραγματεύσεις για το κεφάλαιο 23 και 24 γιατί για μας ε, εδώ θα ήταν ε, θέματα που μας αφορούν ανεξαρτήτως των δικαστικών. Και είναι καλό που παρακολουθείτε την έκθεση προσχώρησης, κύριο Μπιόλης, επομένως θα μπορούσατε να μας βοηθήσετε στο διευρυμένο Προεδρείο όταν θα καταρτήσουμε το πρόγραμμα για φέτο. Για να δούμε πώς μπορούμε, ποια συνέχιση μπορούμε να δώσουμε και πώ μπορούμε να παρακολουθήσουμε την κατάσταση αυτών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία. Τώρα είναι εδώ ο κύριος Μακρύδης, είναι εκπρόσωπος της ε, Κομισιόν. Θα θέλαμε να ακούσουμε και τα δικά σας σχόλια. Συγγνώμη, κοίταξε στη λάθος κατεύθυνση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλησπέρα σε όλους. Και σας ευχαριστώ πολύ που διοργανώνεται αυτή τη συζήτηση που καλύπτει τόσα πολλά ζητήματα, ζητήματα που και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί στενά στη συνεργασία με τις τουρκικές αρχές. Θα ήθελα να εστιαστώ πρώτα σε ζητήματα δικαιοσύνης και θεμελιωδών ελευθεριών και να σας παρουσιάσω την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα θέματα αυτά και ορισμένα από τα ζητήματα που θίξατε. Πρώτα απ' όλα για την υπόθεση πίνω Σελεκ. Σελεκ. Καταδεικνύει κατά την άποψή μου προβλήματα δομικά του δικαστικού συστήματος στην Τουρκία, συμπεριλαμβανομένης και της μακράς διάρκειας των ε, δικών. Το γεγονός ότι πολύ συχνά αλλάζουν οι κατηγορίες ή ανατρέπονται οι δικαστικές αποφάσεις, αλλάζουν οι κατηγορίες κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας ή και η σύνθεση του δικαστηρίου. Εδώ υπάρχει βέβαια και κάτι θετικό σε αυτή την περίπτωση. Στο, οι δικαστές στον πρώτο βαθμό δεν δέχτηκαν την απόφαση του ακυρωτικού δικαστηρίου και μετά η τρίτη περίπτωση ήταν η ολομέλεια του ακυρωτικού δικαστηρίου εδώ, του, του Άρα έχουμε μια περίπτωση στην οποία οι δικαστές προσπάθησαν να επιβεβαιώσουν, να διατρανώσουν την ανεξαρτησία τους. Όπως είπα λοιπόν υπάρχουν δομικά προβλήματα στο ποινικό σύστημα και στο δικαστικό σύστημα της Τουρκίας. Υπάρχουν πολλές παλαιές υποθέσεις που δεν έχουν ακόμα εκδικαστεί. Υπάρχει μεγάλη διάρκεια στην απονομή της δικαιοσύνης και αυτό οδηγεί και σε κράτηση, προφυλάκηση επί μακρό χρονικό διάστημα. Μεγαλύτερη διάρκεια προφυλάξηση από οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα άλλο πρόβλημα είναι οι αποφάσει προφυλάκηση που εκδίδουν τα δικαστήρια. που έχουν δυσμενές αντίκτυπο στα, στο δικαίωμα υπεράσπισης στα δικαιώματα του κατηγορουμένου, καθώς επίσης και η ε, υπονόμευση των δικαιωμάτων στην ελευθερία της έκφρασης και του δικαιώματος του συναθρίζεστε. Συνεργαζόμαστε με τη Δικαστική Ακαδημία, με τους συλλόγους δικαστών και εισαγγελέων προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα αυτά ε, το τρίτο πακέτο μεταρρυθμίσεων έχει εισάγει κάποιες αλλαγές που θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Για παράδειγμα, ε, δικαστές οι οποίοι θα λαμβάνουν αποφάσεις μόνο σε ζητήματα ε, στέρησης της ελευθερίας. Ε, την δυνατότητα άσκησης μάλλον θέσεις του κατηγορημένου με, σε, σε καθεστώς περιοριστικών όρων αντί για προφυλάκηση καθώ επίση και την ανεξαρτησία των εισαγγελέων από το, από το υπόλοιπο δικαστικό σώμα. Ευελπιστούμε αυτές οι μεταρρυθμίσεις να εφαρμοστούν και να εμβαθυνθούν περισσότερο με το τέταρτο πακέτο μεταρρυθμίσεων. Τώρα, σε σχέση με το δικαστικό σώμα, υπάρχει το ζήτημα της ανεξαρτησίας από την εκτελεστική και την ομοθετική εξουσία, αλλά επίσης και το ζήτημα της ανεξαρτησίας των μεμονωμένων δικαστών σε σχέση με την ιεραρχία τους. Δηλαδή δεν πρέπει να δούμε μόνο την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος από τις, τις υπόλοιπες εξουσίας, αλλά και την εσωτερική ανεξαρτησία. Στο πρώτο ζήτημα της ανεξαρτησίας από τις υπόλοιπες, ε, τη διακρίση των εξουσιών. Το 2010, με συνταγματική μεταρρύθμιση, δημιουργήθηκε ένα συμβούλιο που κρίνει ε, την εξέλιξη την επαγγελματική των δικαστών 16 από τα 22 μέλη του οποίου εκλέγονται από τους ομολόγους τους, από άλλους δικαστές. Αυτό θεωρούμε ότι είναι ε, σε ένα σημαντικό βήμα προς την εμπέδωση του κράτους δικαίου στην Τουρκία σε ανταπόκριση των εκκλήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης. λαμβάνεται υπόψη στην επαγγελματική εξέλιξη των δικαστών το κατά πόσον συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των εφετείων και του ανώτατου δικαστηρίου. Αυτό ε, περιόριζε την ανεξαρτησία τους και καταργήθηκε με τις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις του 2010. Άρα από θεσμική άποψη θεωρούμε ότι έχουν γίνει βήματα για την διασφάλιση της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος, αλλά αυτό πρέπει να εφαρμοστεί και στην πράξη. Και όπως ανέφερα, συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με τη Δικαστική Ακαδημία, με το Σώμα των Δικαστών, για να βελτιώσουμε με ε, τα κριτήρια βάσει των οποίων λαμβάνονται οι αποφάσεις για την επαγγελματική εξέλιξη των δικαστών και των εισαγγελέων. Τώρα ένα σχόλιο σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη. Αναφέρθηκε και στο πακέτο διεύρυνσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρυσι. Αν συνεχίσουμε να... Μάλλον. Εάν θέλουμε η Τουρκία να συνεχίσει να προχωράμε τα ρυθμίσεις με βάση την Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση τα απαιτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σημαίνει αυτό ότι πρέπει να υπάρχει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα, σαφές οδικός χάρτης για την ένταξη της Τουρκίας. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας φέτος, πιστεύω. Ευχαριστούμε. Η κυρία Βρεσιά, θέλει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ. Αν τη γνωρίζω ότι δεν συνηθίζεται να λαμβάνει. Να μου λαμβάνω το λόγο τώρα εξεπλάγει λίγο από αυτά που είπατε. Γιατί υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που επανειλημμένα θέτουν οι υπερασπιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία και αυτό είναι ότι οι δικαστέ λαμβάνουν τι αποφάσει του με βάση μόνο το αποδεικτικό υλικό που του παράσχει η αστυνομία χωρί καμία ανεξάρτητη δικαστική έρευνα. Και πιστεύω ότι εκεί υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στην Τουρκία. Δηλαδή, το αστυνομικό έργο σε σχέση με το δικαστικό έργο, με το έργο που θα έπρεπε να γίνεται από τη δικαιοσύνη πλήρως ανεξάρτητα. Σε κάθε περίπτωση εξαρτήτως του πώς λειτουργεί η αστυνομία στην Τουρκία η, η δικαιοσύνη θα έπρεπε να έχει τη δυνατότητα να διεξάγει μια έρευνα πέραν από το αποδεικτικό υλικό που τη παράσχει η αστυνομία και όλα τι μαρτυρίε που έχουμε συλλέξει από τις οργανώσει ανθρωπινών δικαιωμάτων μας δείχνουν ότι αυτό δεν συμβαίνει. Ευχαριστούμε. Νομίζω ότι εδώ ολοκληρώνουμε τη συζήτηση για αυτό το σημείο για την αναφορά της αποστολής μας στην Τουρκία και θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να ε, παραμείνει στην ατζέντα των συζητήσεών μας η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία και θα συνεχίσουμε προφανώς τη συνεργασία μας με την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία με την, ε, ε, καθώς επίσης και με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου. Και τώρα Περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας ε, διάταξη. Στην κατάσταση ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων εν ώψη της αποστολής μιας αντιπροσωπείας της Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη χώρα αυτή. και με την οργανώνουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων από κοινού με την Κοινή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκή Ένωση πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατίας της Μακεδονία. Την συνδιοργανώνουμε λοιπόν αυτή την ε, ε, ακρόαση και βλέπω ότι είναι παρούσα και η πρόεδρος της αποστολής μας. Θα χρησιμοποιώ τον όρο Φύρομ, που είναι ο πολιτικά ορθός. Είχαμε και πέρσι προσπαθήσει να οργανώσουμε κάτι τέτοιο. Δεν τα καταφέραμε. Ευελπιστούμε ότι φέτος θα μπορέσουμε να αποστείλουμε την αντιπροσωπεία μας το Φεβρουάριο. Και πάλι λοιπόν καλώς ήρθατε και επισήμως. Ε, κυρία Χατζημαρκάκη. Είναι ο πρόεδρος της αντιπροσωπείας κοινή κοινοβουλευτική επιτροπή Ευρωπαϊκή Ένωση πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία, τη Μακεδονία. Μια και λοιπόν η αντιπροσωπεία μα θα μεταβεί στη Προ-Γιουκοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία το Φεβρουάριο, είναι φτυχέ το γεγονό ότι θα μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψει τώρα. Από ό,τι βλέπω, Όλοι οι παρευρισκόμενοι γνωρίζετε περισσότερα για το θέμα από ότι εγώ. Έχουμε λάβει την τελευταία έκθεση προόδου που έχει ετοιμάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2012 και εκεί αναφέρεται ότι η χώρα συνεχίζει να πληρεί τα απαιτούμενα πολιτικά κριτήρια για να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα έχει νόημα να συνεχιστούν οι ε, διαταξιακός διάλογος. Ωστόσο, θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα ζητήματα του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης και της πρακτικής εφαρμογής των αρχών αυτών, καθώς επίσης και του διαλόγου μεταξύ των ε, μελών του κυβερνητικού συνασπισμού πρέπει να βελτιωθεί. Ελπίζω να μάθουμε περισσότερα για την κατάσταση στην χώρα αυτή. Πέρα από το ζήτημα της ελευθερίας του τύπου, της του τύπου ένα άλλο θέμα που απασχολεί την Επιτροπή μας είναι η πρόσφατη απόφαση του τμήματος Μίζων σύνθεση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το Δεκέμβριο στην ε, ε, υπόθεση Ελμασρή εναντίον πρώην Ιουκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Συνοπτικά, τι συνέβη σε αυτή την υπόθεση. Ο κύριος Ελμασρή έχει τη γερμανική και την μακεδονική υπηκότητα και στο πλαίσιο του πολέμου κατά της τρομοκρατίας απήχθη στην πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία, με τύχθη στο Αφγανιστάν όπου υπέστη βασανιστήρια το κατηγορούσαν ότι είχε σχέσεις με την Αλκάιντα ή άλλες τρομοκρατικές ομάδες προσέφυγε στα δικαστήρια ε, ένα από τα ε, πράγματα που υπέστη ο κ. Ερμαστή ήταν βασανιστήρια και κακομεταχείριση κατά το χρόνο κράτησή του στην πρώην Ιουκοσλαβική Μακεδονία τη Δημοκρατία. τη Μακεδονία. Ένα άλλο ζήτημα σημαντικό για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή είναι η κατάσταση των Ρωμά. Έχουμε και άλλου προσκεκλημένου για την ανταλλαγή απόψεων, ο κ. Μαρκ Γκρουπερ Διευθυντή τη ε- Ευρωπαϊκή Ομοσπονδια Δημοσιογράφων. Θα, μας, θα αναφερθεί αναλυτικά στο ζήτημα τη ελευθερία του τύπου στη Μακεδονία. Κυρία Χέδερ Κράμπε, διευθύντρια του Open Society European Policy Institute, Ινστιτούτο στι Βρυξέλλε. Έχει συνεργαστεί με τον κύριο Χολιρέν. με την ιδιότητα που είχε ως ε, ε, Επίτροπος για τη Διεύρυνση. Και όπως γνωρίζετε, το Ινστιτούτο Open Society έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα στα Δυτικά Βαλκάνια. Υλοποιεί πολλά έργα ενίσχυσης της εμπλοκής της κοινωνίας των πολιτών στην περιοχή. Έχουμε επίσης από την Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δύο εκπροσώπους, οι κυρίες Σφάικ Πρίστ υπεύθυνη για θέματα διεθνούς πολιτικής και θεωρητικά θα έρθει αργότερα και ο συνάδελφός μας ο κύριος Χάουιτ ο εισηγητής της ΑΦΕΤ, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων για την πρώην Οικοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Και τώρα ίσως κύριε Χατζημαρκάκη θα μπορούσατε να ξεκινήσετε τη συζήτησή μας. Ευχαριστώ κυρία Λόχμπίλερ που μου δώσατε τη δυνατότητα να μιλήσω λίγο για την κατάσταση στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Η έκθεση πρόοδου που έχετε μπροστά σας είναι θετική. Πρέπει να ξέρετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Κοινή Κοινοβουλευτική Επιτροπή πάντα είναι στο πλευρό των ετουσών χωρών, των υποψηφίων χωρών. Προσπαθούμε να είμαστε φίλοι καλοί όλων των χωρών που θέλουν να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η ΦΥΡΟΜ έκανε ιδιαίτερη πρόοδο στους περισσότερους τομείς. Παρ' όλα αυτά υπήρξαν ερωτηματικά σε ορισμένα θέματα. Κάνω λοιπόν καταρχήν μια συνολικά θετική αξιολόγηση λόγω της οικονομικής κρίσης και με δεδομένη την κρίση οι δείκτες της χώρας είναι καλοί, αλλά θέλω να περάσουμε στα ερωτηματικά τώρα. Το πρώτο ερωτηματικό αφορά τις διεθνικές ή διεθνωτικές σχέσεις. Θα γνωρίζετε ότι υπάρχει μεγάλη ε, πλειοψηφία ή μάλλον πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Θα έλεγα ότι η πλειοψηφία της κοινωνίας, των μελών της κοινωνίας, είναι μη αλβανόφωνη και η μεγάλη μειοψηφία είναι ε, ε, αλβανόφωνη και είχαν προβλήματα μετά την ανεξαρτησία της χώρας. Και κατά τη διαδικασία της Αχρίδας, που ανάγεται στη Συμφωνία της Αχρίδας, λύθηκαν κάποια πράγματα, συμφωνήθηκαν, αλλά δεν έχουμε μια κατάσταση λειτουργική όπως στην ε, Ελβετία. Δεν είναι Ελβετία. Υπάρχουν ακόμα προβλήματα που αναφύονται πολλές φορές και άλλες φορές ε, πέφτουν σε, γίνονται λανθάνοντα. Είχαμε το πρώτο εξάμεινο του 2012 κάποια επεισόδια, δολοφονίες στη χώρα που συνέβαλαν στην αύξηση των εντάσεων και των διαμαρτυριών. Ε, η κυβέρνηση αντέδρασε με όριμο τρόπο στις ε, διεθνωτικές αυτές εντάσεις και προσπάθησε να κάνει ό,τι το καλύτερο. Όμως στην κοινωνία όταν γίνονται σκοτομοί μεταξύ των εθνοτήτων αμέσως κλιμακώνονται οι εντάσεις. Ε, μετά θέλω να αναφερθώ στις σχέσεις με τους γείτονες. Ξέρετε ότι η χώρα έχει πρόβλημα με έναν νότιο γείτονα, ε, με τον νότιο γείτονα για το όνομα, αλλά εγώ δεν θα τονίσω αυτό το θέμα εδώ. Εγώ θα τονίσω κάποια προβλήματα που είναι εντονότερα με τον εξανατολών γείτονα, τη Βουλγαρία. Και αυτό είναι κάτι που μας αφορά πάρα πολύ γιατί άπτεται των πολιτικών δικαιωμάτων των πολιτών που έχουν διπλή υπηκότητα ή που ζητούν την βουλγαρική υπηκότητα. Υπήρξαν περιπτώσεις που μας αναφέρθηκαν όπου άνθρωποι που κάνουν, που βάλουν το αίτημα είναι πολίτες της Φύρομ και ζητούν άλλες υπηκότητες, κυρίως τη βουλγαρική και ως ένα βαθμό παρακολουθούνται οι άνθρωποι αυτοί, επικρίνονται και ανοιχτά μάλιστα επικρίνονται. Και θα σας πω ότι στη δική μας ε, μεικτή κοινοβουλευτική επιτροπή έχουμε βουλγάρους ε, συναδέλφους από όλες τις πολιτικές ομάδες και βλέπω μια εξέλιξη εκεί ότι όλοι δηλαδή αναδεικνύουν προβλήματα που δεν υπήρχαν πριν από δύο χρόνια ή δεν αναδεικνύονταν. Ε, γιατί φαίνεται ότι υπήρξαν περιπτώσεις ανθρώπων που επλήγησαν Σπάσκα Βίτρωμα, η υπόθεση Λιζίνσκι, Μαραμπούνεβα που είναι ένα μνημείο το οποίο, στο οποίο επι, επιτέθηκαν ε, ε, βουλγαρικό δηλαδή μνημείο. Αυτά λοιπόν μας τα είπαν οι βουλγαροί συνάδελφοι όλων των κομμάτων και έγιναν συνομιλίες μεταξύ υπουργών, ε, υπουργών εξωτερικών υποθέσεων, αλλά είναι πολύ πιο λεπτό το θέμα τώρα. Υπάρχει ευαισθητοποίηση λόγω της κοινή κληρονομιάς, λόγω της εγκύτητας της γλώσσας, της συγγένειας, της κοινή ιστορίας. Είναι πολύ πιο έντονο το θέμα από ό,τι στη Φύρομ. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι εδώ ο χρόνος κυλά γρήγορα. Ε, οι ελληνικές ανησυχίες μειώνονται κατά τη, όχι πολύ, ενώ οι, βουλγαρικές ανησυχίες για θέματα πολιτικών ελευθεριών επιτείνονται. Είπατε κι εσείς για τους Ρωμά Κάποια πρόοδος υπήρξε στους Ρωμά, γιατί ενέκρινε η κυβέρνηση στρατηγική για να συμπεριλάβει τους Ρωμά, είναι για να καλύψει η στρατηγική το διάστημα 12-14, τη συνοδεύεται με σαφές πρόγραμμα δράσης, το οποίο χαιρετίζουμε εμείς πολύ. Είδαμε όμως παρόλα αυτά ότι υπήρχαν όχι καταχρήσεις, αλλά έγινε χρήση της πολιτικής, της νέας πολιτικής θεωρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιτρέπει στους πολίτες να φύγουν από τη χώρα που οδήγησε σε καταστάσεις όπου η χώρα που εκπροσωπώ σε αυτό το κοινοβούλιο, η Γερμανία, ε, αμφισβήτησε το νέο καθεστώς θεωρήσεων λόγω της εισόδου κυρίως Ρώμα στη Γερμανία. Ε, πολύ μεγάλη εισρωή, πολύ μεγαλύτερη από τα προηγούμενα χρόνια από Φύρομ στη Γερμανία. Και αυτό δείχνει ότι η στρατηγική αυτή τη συμπερίληψη χωρίς αποκλεισμούς δεν λειτουργεί πάντα πολύ καλά, τέλος πάντων μπορεί να βελτιωθεί. Θέλω να αναφέρω κάποια επεισόδια που αφορούν τα μέσα ενημέρωση και ο κύριος Γκρούμπερ θα μιλήσει για αυτά, αλλά μπορούμε να πούμε ότι εμεί ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με τον Επίτροπο Φίλε που είναι μάλιστα τώρα στα Σκόπια ε, έχουμε ξεκαθαρίσει το θέμα της ελευθερίας των ΜΜΕ διότι υπήρξαν πολλά παραδείγματα όπου παρενέβη η κυβέρνηση εντονότατα και υπήρξε έντονη αντίδραση καθόλου διπλωματική, <laughs> καθόλου χαρακτηριστική από τον Επίτροπο Φίλε. Οπότε και εμείς στο Κοινοβούλιο πρέπει να παίξουμε το ρόλο του καλοπροαίρετου διαπραγματευτή, γιατί η ένταση ενάντια στην Επιτροπή κλιμακώθηκε. Πάντως όλα αυτά οδήγησαν σε ένα στρογγυλό τραπέζι από τον Τεού Ταρίφη, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρέπει... Α, η κυρία είναι. Σε τεχνική βάση μπόρεσε να ε, ε, φέρει όλα τα μέρη σε ένα στρογγυλό τραπέζι και αυτή η διαδικασία βοήθησε πάρα πολύ από την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και οδήγησε σε βελτίωση της κατάστασης μέχρι ότου πολύ πρόσφατα στις 24 Δεκεμβρίου δυστυχώς κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικής συνόδου για τον προϋπολογισμό το μεγαλύτερο ε, κόμμα της αντιπολίτευσης, οι σοσιαλδημοκράτες προκάλεσαν επεισόδιο μέσα στο κοινοβούλιο μετα, ε, προσήχθησαν βιαίως εκτός του Κοινοβουλίου έχει γίνει και εδώ κατά το παρελθόν αλλά εν προκειμένου πολλούς τους έβγαλαν έξω οι ε, υπεύθυνοι για την ασφάλεια εξεδιώχθησαν και δημοσιογράφοι από το Κοινοβούλιο και από τότε κάνουν μποϊκοτάζ ε, στο Κοινοβούλιο η αντιπολίτευση και αυτό είναι ένα βήμα πίσω. Οπισθοδρόμηση. Πρέπει λοιπόν εδώ ξεκάθαρα εμείς να μιλήσουμε για αυτό το θέμα σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο κύριος Κάμερα, ο συνάδελφος από την Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή είναι εδώ και πρέπει να αποφασίσουμε πώς θα γίνει μια επίσκεψη Ω Μεικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή στη χώρα στις αρχές Φεβρουαρίου. Γιατί έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα δεν μπορούμε να πάμε εκεί. Περιμένουμε να μας δοθούν σαφή δείγματα γραφής. Αύριο θα κάνουμε μια συνάντηση για να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε, διότι ένα κοινοβούλιο ε, το οποίο τον μποϊκοτάρουν δεν μπορούμε εμεί να το επισκεφτούμε μίλησα με τον Υπουργό Εξωτερικό χθε. Θέλουμε να βρούμε μια λύση, ούτω ώστε τα μέρη να προσεγγίσουν πάλι. Να βοηθήσουμε κι εμεί. Αλλά η τωρινή κατάσταση σαφώ είναι δυσχερέστατη. Η... Το δικαίωμα του συναθρίζεστε είναι δεδομένα. Δεν ε, ε, υπάρχουν καταχρήσεις εδώ. Για να τελειώνω και του συνέρχεστε είναι και αυτό εντάξει. Υπήρξαν περιπτώσεις που υπονομεύθηκαν από το απρόβλεπτο πολιτικό τοπίο. Η καλή, η θετική πρόοδος ισχύει ε, για τους περισσότερους τομείς που καλύπτονται από διαπραγματευτικά κεφάλαια, το κεφάλαιο 23, το 24, ασφάλεια, ε, ελευθερία τη δικαιοσύνη του 23, αλλά με τις πρόσφατες εξελίξεις κατά νουν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να ασκήσουμε πιέσεις που έπαιξαν ρόλο θετικό, ανέφερα τον κύριο Φίλε, και τις δικές μας ενέργειες. Πρέπει να ασκήσουμε πίεση λοιπόν, ώστε η χώρα να παραμείνει στο σωστό δρόμο. Γιατί εμείς θέλουμε να αρχίσουν διαπραγματεύσεις το, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το θέλει αυτό, αλλά δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μας μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Χατζημαρκάκη και σας ευχαριστούμε που αναφερθήκατε και στο ότι η αντιπροσωπεία σας μπορεί να αποφασίσει υπέρ ή κατά της επίσκεψης αύριο. Έχουμε ένα διευρυμένο προεδρείο και θα το συστήσουμε και αυτό το θέμα. Αλλά επειδή έχουμε την έκθεση μόλις για την αποστολή στην Τουρκία, υπάρχει μια ομάδα βουλευτών που μποϊκοτάρουν το Κοινοβούλιο. Για μας αυτός δεν είναι ο λόγο που δεν θα πρέπει να συζητήσουμε την κατάσταση των ανθρωπινών δικαιωμάτων, αλλά θα είμαστε σε επικοινωνία για το τι θα αποφασίσουμε. Ο επόμενο ομιλητή, ο κ. Γκρούμπερ, είναι ο διευθυντή τη Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε καθώς ε, ε, μιλάμε για πολυγλωσία, θα μιλήσω γαλλικά στη μητρική μου γλώσσα. Έρχεται σε μια πολύ χρήσιμη χρονική στιγμή η συζήτηση αυτή, γιατί το θέμα της ελευθερίας του τύπου εδώ και χρόνια συζητείται μεταξύ των δημοσιογράφων ε, στη Φιρόμ, αλλά η κατάσταση εντυπωσιοποιήθηκε κάπως τους τελευταίους μήνες. Καταρχήν τον Νοέμβριο είχαμε την υιοθέτηση ενός νόμου για την αποποινικοποίηση ε, των αδικημάτων της δυσφήμισης και της συκοφαντία κάτι που αναμενόταν ιδιαίτερα από τους δημοσιογράφους ε, και έθεσε τέλος ε, σε 700 υποθέσεις ε, κατά των δημοσιογράφων της, στην, ε, και θα λέω Μακεδονία Λεωμιλητής για να μην ακρηγορώ. Όπως ε, είπε και ο κύριος Χατζημακάκης, το Δεκέμβριο είχαμε ένα περιστατικό στο Κοινοβούλιο, μια ομάδα δημοσιογράφων εκδιώχθηκε βία από τα σώματα ασφαλείας του Κοινοβουλίου και θυμάμαι ότι σε αυτό το πλαίσιο προχτές η ομάδα υψηλού επίπεδου για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, που συστέθηκε από την κυρία Κρούς ανέφερε μεταξύ των συστάσεων ότι κάθε έτοιμο προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διέπεται από κριτηρία ελευθερίας του τύπου ε, πάρα πολύ αυστηρά. Δηλαδή στην περίπτωση που δεν ήταν ε, ξεκάθαρα τα πράγματα, τουλάχιστον τα ξεκαθάρισε αυτή η ομάδα, γιατί για να υπενθυμίσω κάτι που είχαμε πει από το 2004, ε, αυτό δεν είχε υποθεί σαφώς. Για να επανέλθω τώρα στο ζήτημα, στην ουσία του ζητήματος. Ε, η κατάσταση της ελευθερίας των ΜΜΕ στην Δημοκρατία της Μακεδονίας είναι, όπως είπε ο κ. Χατζημαρκάκης, είτε στο ζεστό είτε στο κρύο. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες πρόοδοι, αλλά ξεκολουθούν να υπάρχουν πολλά προβλήματα. Παραδείγματο χάρη το πολιτικό και το νομικό περιβάλλον ε, που δεν ωφελούν ιδιαίτερα την ελευθερία έκφραση των δημοσιογράφων. Υπάρχει πάρα πολύ αυτολογοκρισία και κάποιες οικονομικές ε, συναλλαγές που δεν γίνονται σε απόλυτη διαφάνεια και επίσης κάποια γεγονότα που ε, αναφέρω, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που ξεχνάμε όταν ε, μιλάμε για την ελευθερία της έκφρασης, για την καθημερινή δουλειά των δημοσιογράφων. Μιλήσαμε για την ελευθερία του συνέρχεστε. Έχουμε τέσσερι συγκεκριμένε περιπτώσει δημοσιογράφων που έχουν ε, ε, προσληφθεί από τα μέσα στην Μακεδονία και τους ζητήθηκε να υπογράψουν ένα προληπτικό, μια προληπτική επιστολή για να εγκαταλείψουν το συνδικάτο τους ή για να εγκαταλείψουν τη θέση της εργασίας τους αν κάποια στιγμή κάτι έλεγαν που δεν άρεσε σε κάποια πρόσωπα. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό μέσο πίεση ε, κατά την άποψή μας ε, και μάλιστα το αναφέραμε στον Επίτροπο Φίλε. Υπάρχει λοιπόν πίεση σε όσους θέλουν να ε, συμμετέχουν στα συνδικάτα, στην ΦΥΡΟΜ και ουσιαστικά δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις, ασκούν πάρα πολύ μεγάλη πίεση οι εργοδότες και όσοι ελέγχουν τα μίντια. Αυτό σε ό,τι αφορά τι συνθήκε εργασία. Όπω αναφέρθηκε προηγουμένω, πράγματι υπάρχουν κάποιε περιπτώσει στο παρελθόν, κάποιε εταιρείε μέσω ενημέρωση ήταν αντικείμενο αποφάσεων αυθαίρετων κατά την άποψή μα ή τουλάχιστον αμφισβητήσιμων ή σκοτεινών. Ε, μιλώ, παραδείγματο χάρη, για την τηλεόραση ΕΤΒΕ που έκλεισε ε, και δεν έχει γίνει αυτή η διαδικασία σε, δια, σε διαφανείς διαδικασίες. Έχασε την αδειά της ε, η εταιρεία ή έκλεισε για λόγους φόρο αποφυγής ενώ καμία έρευνα δεν είχε γίνει για άλλα μέσα που θα μπορούσαν να είναι στην διακατάσταση. όπως ε, καθώς συστήθηκε ένας διάλογος μεταξύ δημοσιογράφων και κυβέρνησης για τη μεταρρύθμιση των ε, μέσων ε, ο διάλογος αυτός ξεκίνησε από τη στιγμή της εκδίωξης των δημοσιογράφων από το Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή παρουσ... προετοιμάζει μία μεταρρύθμιση η κυβέρνηση ε, για το νόμο για τα μέσα, όμως ε, κανείς δεν μπορεί να συζητήσει από τον κλάδο γιατί οι δημοσιογράφοι αρνούνται να συζητήσουν με την κυβέρνηση στις σημερινές συνθήκες. Αυτό είναι και πάλι κάτι ανησυχητικό γιατί κάθε νομοθετική ή πολιτική μεταρρύθμιση δύσκολα μπορεί να γίνει χωρίς ε, τους αρμοδίους του κλάδου, δηλαδή τους δημοσιογράφους και χωρίς τα ίδια τα μέσα. Μίλησα για την τηλεόραση Α1, θα μπορούσα να αναφερθώ και σε μια σειρά εκπομπών που υπάρχουν και είναι διαθέσιμες και αρνούνται τα κανάλια της τηλεόρασης να τις αναμεταδώσουν. Ε, έχω κάποια παράδειγματα, κάποιοι παραγωγοί, παραδείγματος χάρη δημοσιογράφοι, έχουν ε, έτοιμες εκπομπές και κανένα κανάλι τηλεοπτικό δεν τις μεταδίδει. Μπορούμε να μαντέψουμε ότι πρόκειται για πολιτικούς λόγους. Από την άλλη, θα μπορούσαμε τη, να αξιολογήσουμε τη λειτουργία της ε, αγοράς των μέσων ως κάτι αδιαφανές. Ε, γιατί πολλές φορές οι εταιρείε πουλούν, ξαναγοράζουν, κανείς δεν ξέρει σε ποιον ανήκει Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το υπενθυμίσουμε. Δηλαδή, ένα από τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να υπάρχει ένα βαθμό διαφάνεια και μάλιστα πολύ διαφάνεια για την ιδιοκτησία των ε, ΜΜΕ και αυτό λείπει στη χώρα αυτή. Νομίζω ότι όταν διαβάζει κάποιο μια εφημερίδα ή βλέπει τηλεόραση σε συγκεκριμένο κανάλι, θέλει να ξέρει σε ποιον ανήκει, ποιο τον ελέγχει. Υπάρχουν λοιπόν διάφορε καταστάσεις και αυτό μας οδηγεί μακροπρόθεσμα ε, στο εξής μήνυμα ότι για μία χώρα που καθορίζει την ελευθερία του τύπου μία από τις πέντε προτεραιότητε για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι πρέπει να γίνει ακόμη πολύ μεγάλη πρόοδο. Και φυσικά όλα αυτά δεν αφορούν ε, μόνο κάποια κριτήρια την υιοθέτηση ενό νομοσχεδίου, αλλά το σύνολο τη κατάσταση. Δεν είναι καθόλου ικανοποιητικά τα μηνύματα που δεχόμαστε και βλέπουμε ότι απλώς μας πετούν στάχτη στα μάτια και πρέπει να γίνει πολύ μεγάλη πρόοδος για την ελευθερία του που Θα σταματήσω εδώ και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κυρία Γκρούμπα. Και τώρα η κυρία Γκράμπ έχει το λόγο. Uh, ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα εστιαστώ πρώτα απ' όλα στην κατάσταση των Ρωμά, στην οποία αναφέρθηκε και ο κύριος Χατζημαρκάτης, και κυρίως και επίσης στην υπόθεση Αλμασρή. Είναι δύο ζητήματα για τα οποία το Open Society Foundation εργάστηκε. Επομένω, έχω πολλέ πληροφορίε που θα μπορούσα να σα ε, δώσω και ορισμένα ερωτήματα που θα μπορούσα να θέσει η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν επισκεφθεί τη χώρα και κατόπιν ορισμένε άλλε μικρότερε ε, σε διάρκεια παρατηρήσει για την ε, εμπλοκή τη κοινωνία των πολιτών και την κοινοβουλευτική δημοκρατία στην ΦΥΡΟΜ, καθώ επίση και το πρόγραμμα Σκόπια 2014. Πρώτον, για την κατάσταση των Ρωμά. Όπω ανέφερε και ο κ. Χατζημαρκάκη, έχει διατυπωθεί ένα σχέδιο δράση και μια στρατηγική για την καταπολέμηση του αποκλεισμού των Ρωμά. Παρ' όλα αυτά, ο προπολογισμό και τα κονδύλια είναι πολύ μικρά. Πολύ χαμηλή η χρηματοδότηση. Επομένω, θα ήθελα να επισημάνω στην υποεπιτροπή σα Θα ήθελα να προτείνω λοιπόν στην Υποεπιτροπή να τεθεί το ερώτημα στις αρχές της ΦΥΡΟΜ γιατί έχουν ε, δίνονται τόσο ε, μικρά κονδύλια για την αντιμετώπιση του αποκλεισμού των Ρωμά, κυρίω για το ζήτημα της εκπαίδευση, της πρόσβασης στην εκπαίδευση, που είναι εξαιρετικά σημαντικό. Το δεύτερο άλλο σημαντικό ζήτημα είναι πώς η κυβέρνηση ε, επιθυμεί να υλοποιήσει το δεύτερο επιχειρησιακό σχέδιο για τους Ρωμά. Πολύ συχνά αναφέρονται στην, στον αριθμό Ρωμά που συμμετέχουν που εκπροσωπούνται στην κυβέρνηση μέσω ενός Υπουργού Ανευχατοφυλακίου μέσω του Υπουργού Εργασία. Παρ' όλα αυτά, στην δημόσια διοίκηση οι Ρωμά υποεκπροσωπούνται. Είναι εξαιρετικά μικρό ο αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων Ρωμά. Και όλα αυτά τα ζητήματα εξάλλου είχαν αναφερθεί ως περιοχές εστίασης τη δεκαετία για την καταπολέμηση του υποκλεισμού το Ρωμά, ζητήματα που αφορούν στην, ε, στις περιουσίες και η πρόεδρος είναι πολύ μικρή. Ένα από τα συμπτώματα αυτής της αναποτελεσματικής πολιτικής ε, καταπολέμησης του αποκλεισμού των Ρωμά είναι το γεγονό ότι όλο και περισσότεροι Ρωμά κάνουν αιτήσει ασύλου, χωρίς πολιτικού ασύλου, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό έχει και σημαντικές επιπτώσεις στην ίδια τη χώρα. Έχει αυξηθεί η χρήση των ε, φιλετικών χαρακτηριστικών από τους συνοριοφύλακε της δημόρφους εικόνες με βάση αυτά, και υπάρχουν ήδη τρεις σχετικές υποθέσεις εκκρεμής στα εθνικά δικαστήρια. Έχουν καταγγελθεί επίσης, έχει καταγγελθεί επίσης κατα, κακομεταχείριση των Ρωμά. Αυτός ο στιγματισμός αυτής της, της, της ε, μειονότητας έχει οδηγήσει σε ένα φαύλο κύκλο. Ακόμα μία ομάδα η οποία υφίσταται ε, διακρίσεις στην ΦΥΡΟΜ είναι οι ε, λεσβείες, ομοφιλόφιλοι, αμφιφιλόφιλοι και τραξισεξουαλικοί. Η κοινότητα αυτή έχει εκφράσει τα αιτήματά της με μια έκκληση στην οποία δεν ανταποκρίθηκε η κυβέρνηση της ΦΥΡΟΜ. Τώρα θα περάσω στην υπόθεση Ελμασρή. Το Ίδρυμά μας είναι πλάκι άμεσα στην εκδίκαση αυτή τη υπόθεση ε, στην νομική συνδρομή. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε ότι η ΕΣΔΑ παραβιάστηκε σε διάφορα. πολλά άρθρα της παραβιάστηκαν, πρώτον όσον αφορά την απαγόρευση των βασανιστήριων, την ε, παράνομη κράτηση και την παράλευση διεξαγωγή έρευνα το, η κυβέρνηση δεν έχει λάβει τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να ελέγξει τις υπηρεσίες πληροφοριών, να καταργήσει τις, τα παράνομα μυστικά κέντρα κράτηση, καθώς επίσης και να πάυσει να παράσχει ψευδείς πληροφορίες σε διεθνείς οργανισμούς ή υπόθεση πολίτες Πιστεύω ότι η υπόθεση Ελμάστρη είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των προβλημάτων του δικαστικού συστήματο στην Φιρόμ πολλά παραποιημένα αποδεικτικά στοιχεία από τις μακεδονικές αρχές παρασχέθηκαν σε ευρωπαϊκές ε, ευρωπαϊκά όργανα. Χρειάζεται λοιπόν να αντιμετωπιστούν τα δομικά προβλήματα τα οποία επέτρεψαν και δημιούργησαν το πρόσφορο έδαφος έτσι ώστε να υποστεί αυτά τα βασανιστήρια για την μεταχείριση του κ. Ελμάστρη. Επίσης η κυβέρνηση θα πρέπει να ελέγξει τη λειτουργία της ε, υπηρεσίας πληροφοριών, των μυστικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να προλάβει τέτοιες καταστάσεις και να μην επαναληφθούν ποτέ στο, στο, μέλλον. Θα ήθελα λοιπόν η, Υποτροπή, η Υποεπιτροπή και η Αποστολή σας να θέσει το ζήτημα πώς ελέγχεται η λειτουργία των μυστικών υπηρεσιών. Σίγουρα σε είμαι βέβαιη μάλλον ότι θα σας δοθούν ε, επιχειρήματα του τύπου ε, ότι η προηγούμενη κυβέρνηση ε, υφίστατο πιέσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες επειδή επιθυμούσε να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ η χώρα κτλ. Αλλά υπάρχουν συστηματικά δομικά προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν και τα οποία πρέπει θα ενθαρρύνω να θίξετε στις επαφές σας. Γιατί αυτά τα προβλήματα του δικαστικού συστήματος αφορούν και σε υποθέσεις παράνομης λειτουργίας των υπηρεσιών ασφαλείας και των υπηρεσιών, των μυστικών υπηρεσιών και δημιουργούν ένα περιβάλλον ιδιαίτερα επικίνδυνο για τη δημοκρατία. Τώρα, σε σχέση με την κατάσταση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας μετά τα γεγονότα της 24ης Δεκεμβρίου 2012 είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι. Ε, πολλοί ακτιβιστέ, δημοσιογράφοι ή οποιοδήποτε έχει ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση έχει ε, υποστεί διώξει με βάση τον νόμο περί κάθαρσης και το ζήτημα αυτό ετέθη στον υψηλού επίπεδου προενταξιακό διάλογο. Και καλωσορίζουμε αυτήν, αυτό το γεγονό, αλλά θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το θέσει με μεγαλύτερη ένταση στην προενταξιακή διαδικασία. Και τώρα για το πρόγραμμα Σκόπια 2014 θα είχε νόημα ίσω να θέσετε ορισμένα ερωτήματα σε σχέση με τον προπολογισμό, γιατί δεν υπάρχει καθόλου διαφανή διαχείριση των κονδυλίων. Η νομοθεσία για τα δημόσιε δαπάνε τροποποιήθηκε ακριβώ προκειμένου να περιοριστεί και να μειωθεί η εποπτεία. Κονδύλια τα οποία πρόκειται να δοθούν σε δήμου ή κοινότητε οι οποίε δεν πρόσκειται θετικά προ την κυβέρνηση ε, μεταφέρονται αλλού. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κυρία Γκράμπερ για αυτές τις, ε, αυτή τη λεπτομεριακή παρουσίαση. Νομίζουμε ότι θα μας βοηθήσουν τα θέματα που θίξατε να προετοιμαστούμε για την συνάντησή μας. Νομίζω ότι τα ζητήματα που θίξατε για την υπόθεση Ελμάσρη συνδέονται και με τη δεύτερη έκθεση που θα εκδώσει το Κοινοβούλιο σε σχέση με τα μυστικά κέντρα κράτηση και τι εκνομε μεταγωγέ. Δυστυχώ πολλά κράτη δεν παρακολούθησαν την εξέλιξη αυτή τη διαδικασία. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην εκπρόσωπο τη Γενική Διεύθυνση Διεύρυνση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αντί να επαναλάβω αυτά που ελέγχθησαν ήδη από τους ομιλητές που είναι πολλά και διάφορα και σας ευχαριστώ γι' αυτό Επιθυμώ να συμπληρώσω με στοιχεία από άλλους τομείς από τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γενική παρατήρηση καταρχήν. Όλη η χώρα τώρα είναι σε φάση εξέλιξη στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πράγμα αναμενόμενο σε αυτό το στάδιο της διεύρυνσης. Σε κάποιους τομείς, σε κάποιους τεχνικούς, λιγότερο πολιτικούς τομεί έχουν προχωρήσει περισσότερο ίσως τα ανθρώπινα δικαιώματα γενικά είναι ένα τομέα που χρειάζεται χρόνο, πολιτική βούληση, συνεχή κατανομή πόρων οικονομικών από τον προπολογισμό, πραγματογνωμοσύνη και βοήθεια από το εξωτερικό. Καμιά φορά η πρόοδο μπορεί να είναι βραδία και γι' αυτό στην τελευταία έκθεση πρόοδου της Κομισιόν παρατηρήσαμε μια μέτρια ανάπτυξη σε κάποιους τομείς ε, στα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, στα δικαιώματα των γυναικών, των παιδιών, των ανθρώπων με αναπηρίες κλπ. Ακούσαμε για πολλά κενά και προβλήματα μέχρι τώρα, αλλά θα ήθελα και εγώ να σας υποδείξω μια καλή εξέλιξη. Ε, καμιά φορά μπορεί να είναι ασυντόνιστες οι προσπάθειες ε, στα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά εδώ θέλω να μιλήσω καλά για τον διαμεσολαβητή και το γραφείο του που λειτουργεί 15 χρόνια και κάνει έκθεση πάρα πολύ καλή κάθε χρόνο και παίζει ουσιώδη ρόλο γιατί προστατεύει τους πολίτες και τα δικαιώματά τους απέναντι στα κρατικές υπηρεσίες και τώρα κάνει και εκστρατείες ευαισθητοποίησης και προσέχει ιδιαίτερα τα δικαιώματα των παιδιών, έχει ειδικό τμήμα για τα δικαιώματα των παιδιών και την πρόθεσή τους και την αντιμετώπιση κρατουμένων φυλακισμένων. Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα λοιπόν για την περιοχή που πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, να το έχετε και εσείς που θα πάτε εκεί. Ε, έχω επιλέξει κάποιους τομείς ε, που προκαλούν κάποιες ανησυχίες ε, και δεν αναφέρθηκαν μέχρι τώρα από τους ομιλητές. Η Κομισιόν επανειλημμένα εξέφρασε ανησυχία για την κατάσταση στη, στα κρατητήρια και τις φυλακές, ιδιαίτερα την φυλακή Ρίζη. Η Επιτροπή Πρόληψη Βασανιστήριων του Συμβουλίου της Ευρώπης ασχολήθηκε με αυτό το θέμα και μέσα του περασμένου μήνα έκανε μια διεξοδικότατη έκθεση σχετικά. Επίση επιβεβαιώνονται οι ανησυχίε μας από το ίδιο το Γραφείο του Εθνικού Διαμεσολαβητή, ο οποίος κάνει επιθεωρήσει πολύ συχνά με το ρόλο του ως ε, ε, οργάνου και μέσου πρόληψης ε, στα πλαίσια του προγράμματος ΟΠΚΑΤ. Επίσης υπάρχουν προβλήματα υγιεινής, τροφίμων, ε, κακής υποδομής, κακής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, συνοστισμός, βία μεταξύ των φυλακισμένων, ανεπαρκείς φύλακες σε σχέση με το πληθυσμό των κρατουμένων κλπ. Έχουν γίνει κάποια μικρά βήματα μπροστά και τα κρατάμε, για παράδειγμα βελτιωμένη ε, κατάρτιση και διαδικασίες. Ε, την περασμένη άνοιξη η αποστολή μας ανέφερε καταχρηστικές συμπεριφορές από φύλακες των φυλακών και ε, μειώθηκε, μειώθηκε η ε, καταχρηστική πρακτική και η απομόνωση. Αλλά όμως διαφθορά παραμένουν. Επίσης ε, υπάρχει ένα μεγάλο πρόγραμμα το οποίο θα δημιουργήσει καινούργιες πτέρυγες των φυλακών για να μειωθεί ο συνοστισμός. Αυτό όμως είναι μόνο μέρος της λύσης παραμένει το θέμα του δημοσιονομικού, λίγη πόρη από τον προϋπολογισμό, ε, λίγο προσωπικό, αυτά δημιουργούν προβλήματα. Ε, ένα άλλο θέμα που αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες που δεν το αναφέραμε είναι το δικαίωμα για δίκαιη δίκαιη από αμερόληπτο ανεξάρτητο δικαστήριο μέσα σε έφθετο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι σημαντικό μεταξύ 4 και 5 χιλιάδες προσφυγές που χειρίζεται ο Εθνικός Διαμεσολαβητής Ετησίως. Από αυτές το μεγαλύτερο κομμάτι έχει να κάνει με τη δικαστική εξουσία και εδώ είναι η διάρκεια της διαδικασίας. Το Υπουργείο η δικαιοσύνη στο ανώτατο δικαστήριο επίσης ε, παραλαμβάνει κάθε χρόνο πολλές αναφορές για τα προβλήματα αυτά της ε, ε, μακράς διάρκειας και τη συμφόρησης της υποθέσεις που εκκρεμούν και εδώ υπάρχουν και πολλές ε, παραβιάσεις. Ε, τώρα έχουν γίνει κάποια βήματα για να εξυγχρονιστεί το σύστημα της δικαιοσύνης. Ε, υπάρχουν πολλές ε, βελτιώσεις σε σχέση με τις ε, δίκες που εκκρεμούν. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να στοχευθούν και να επιληθούν υποθέσεις που δεν εκδικάστηκαν. Ε, είναι πολύ δύσκολο να εξευρεθούν γιατί δεν έχουμε πολλές φορές λεπτομέρειες για να τις βρούμε. Τώρα, για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Πάλι εδώ υπάρχουν υπέρ και κατά. Στα υπέρ η νομοθεσία υπάρχει νόμος που έχει ευθυγραμμιστεί με το κεκτημένο και όλες τις διεθνείς νόρμες, με μία εξαίρεση ναι, το σεξουαλικό προσανατολισμό που είναι λόγος διάκρισης εκεί στη χώρα αυτή και η Επιτροπή Καταπολέμησης των Διακρίσεων λειτουργεί τα τελευταία δύο χρόνια όμως ο διαμεσολαβητής ε, θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει βελτιωμένη, είναι πολύ χαμηλή η ευαισθητοποίηση. Επίσης η Επιτροπή και ο διαμεσολαβητής στην πράξη χειρίζονται θέματα που αφορούν τους ΛΟΑΔ, βίες, ομοφυλόφους κλπ. Δεν υπάρχει μεγάλη παρουσία εκπροσώπων από αυτές τις ομάδες. Η ευαισθητοποίηση είναι πολύ χαμηλή και αυτό είναι από τα πιο παραμελημένα θέματα στη χώρα. Ένα τομέα όπου θα επικαλυφθώ με του προηγούμενου ομιλητέ είναι η ελευθερία έκφραση που κυριάρχησε στην ημερήσια διάταξη πέρσι στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θυμίζω τις επιτυχίες από αυτή την ιστορία. Το Νοέμβριο άρθρα από τον ποινικό κώδικα που αφορούν τη συγκοφαντική δυσφήμιση έχουν ανακληθεί και εγκρίθηκε πολιτικός κώδικας σε συμφωνία με το άρθρο 10 της Σύμβασης για ε, την Ελευθερία Έκφρασης από ποινικοποίηση της ε, συκοφαντικής δυσφήμισης ε, είχε προωθηθεί από το ε, ΝΟΑΣΕ, το Υγνοπληκτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης και τον δικό μας τον Επίτροπο. Η χώρα λοιπόν έκανε μια μεταρρύθμιση όπου η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του Συμβουλίου τη Ευρώπη, δεν έχουν ακόμα κάνει. Οπότε αυτό είναι πολύ μεγάλο βήμα, αλλά είναι το πρώτο βήμα και πολλά θα εξαρτηθούν από την πρακτική εφαρμογή τη Νέα νομοθεσία και την ερμηνεία του από τα δικαστήρια. Θα δούμε. Τελευταίο σημείο, τι έγινε στις 24 Δεκεμβρίου στο Κοινοβούλιο, αυτό δημιούργησε, έκανε ζημιά και είναι ε, κακό γιατί έρχεται σε άσχημη στιγμή μετά τα καλά σχόλια ε, και τις καλές επιδόσεις από πέρσι, όπως είπε και ο κύριος Χατζημαρκάκης. Ε, η ομάδα εργασίας για τα μέσα ήταν καλό φόρουμ, έδωσε αποτελέσματα, δούλεψε καλά. Ήταν ένα βήμα για, ώστε η Ένωση Δημοσιογράφων να παρακαθίσουν μαζί με την κυβέρνηση και να λύσουν προβλήματα μέσα από το διάλογο και τους ενθαρρύνουμε και τους καλούμε να επιστρέψουν στο διάλογο. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για την αποποινικοποίηση τη συμφωνική της αλλά και τα εργασιακά δικαιώματα των δημοσιογράφων, ε, αυτορύθμιση από τους δημοσιογράφους, βελτίωση των κωδικών δεοντολογίας κλπ. Οπότε ακόμα αυτό το φόρουμ για τα ΜΜΕ πολλά έχει να κάνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και νομίζω ότι τώρα έχουμε μια πλήρη εικόνα με όλες τις παρουσιάσεις ε, μπορούμε να κατανοήσουμε πού σημειώθηκε και πού δεν σημειώθηκε πρόοδος, ε, ακόμη και μάλιστα που επιδεινώθηκε η κατάσταση. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε και το χρόνο κατά νου. Έχουμε τον κύριο Κούκα στον κατάλογο των ανθρώπων που ζητήσει το λόγο. Ποιος άλλος από τους συναδέλφους, ο κύριος Κράμερ και η κυρία Γιάννα Κουδάκη. Ο κύριος Κούκαμ. Ευχαριστώ. είμαι σύντομο γιατί όλα τα θέματα που ήθελα να αναφέρω εγώ αναφέρθηκαν από του προλαλήσαντε. Ιδίω από τον κύριο Χατζημαρκάκη μας παρουσίασε μία πλήρη εικόνα τη κατάσταση στη χώρα. Αναφέρω το θέμα της ισότητα των δύο φύλων δεν ε, ε, υπάρχει στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στην αγορά εργασίας η διάσταση αυτή. Και μάλιστα όμως πρέπει να σας πω ότι σε σχέση με τα περισσοτερα κρατημέλη, σε ό,τι φορά ε, τους βουλευτές έχει πάρα πολύ υψηλό ποσοστό η πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, αλλά θα πρέπει ε, ουσιαστικά στην πράξη να προωθηθούν και να διαφυλάσσονται τα, πρόσθετα, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης ε, πρέπει να ενδυναμωθεί η διοργανική συνεργασία, η διοικητική ικανότητα και να υπάρξει ευαισθητοποίηση, οικοδόμηση εμπιστοσύνη μεταξύ των κοινοτήτων. Είναι ένα από τα καθήκοντα της χώρας για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μία ακόμη παρατήρηση, όπως ε, και να δούμε την κατάσταση. Εγώ δεν πιστεύω ότι να εμποκοτάρουμε το Κοινοβούλιο είναι ο σωστός ε, τρόπος να πετύχουμε πολιτικά αποτελέσματα. Θα πρέπει να γίνουν όλα αυτά εντός του Κοινοβουλίου. Όποια και αν είναι η ευριανή σας απόφαση για το να μεταβούμε ή όχι εκεί, Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δείξει μεγάλη ευαισθητοποίηση απέναντι στη δική σας απόφαση, δηλαδή να αποφευχθεί η πιθανή ερμηνεία ότι αν δεν μεταβούμε εκεί, αν δεν μεταβείτε εκεί, εσείς ενθαρρύνετε τις πολιτικές δυνάμεις που μπλοκάρουν την τακτική λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών σας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Κούκεν. Ο κύριος Κράμερ. Ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις. Πριν από δύο χρόνια ε, κάναμε συζήτηση στα Σκόπια για να δούμε αν η Μακεδονία πληρεί το, και θα υιοθετήσει το χάρτη για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τον ε, υιοθέτησαν το χάρτη, αλλά έβγαλαν το κομμάτι που αφορά τον σεξουαλικό προσανατολισμό για να μην αναγνωρίσουν την ομοφιλοφιλία. Τα συζητήσαμε αυτά, δεν έχουμε προβλήματα. Όμως, ένα είναι σαφέ, είπα ότι αν δεν το υιοθετήσουν και αυτό, δεν μπορούν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. άλλα δεν τους ενδιαφέρει, ε, αυτό όμω δεν ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει η Κομισιόν πώ αντέδρασε τι αντιδράσει υπήρξαν μετά τι εξελίξεις. Ε, ακούσαμε ότι επιδεινώθηκαν τα πράγματα και δεν βελτιώθηκαν. Τέλος, είτε πάμε είτε δεν πάμε, Πρέπει να πω ότι το ταξίδι της αντιπροσωπείας έπρεπε να είχε γίνει πριν από δύο μήνες. Και είχαμε κάνει και τις κρατήσεις μας, ή μεγάλο κομμάτι των βουλευτών, μεγάλη μερίδα έκαναν κρατήσεις και τα πήραν πίσω γιατί ο πρόεδρος της αντιπροσωπείας ασθένησε. Και αυτό ανθρώπινο είναι, αλλά υπάρχουν αναπληρωτές, ξέρετε, για κάθε αξίωμα. Αλλά επειδή όμως αναπληρωτής ήταν από άλλο κόμμα, ε, φραναρίστηκε και ακυρώθηκε το ταξίδι. Ανεξάρτητα με το τι κάναμε εμεί. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να ε, μεταχειριζόμαστε έτσι την αντιπροσωπεία. Εγώ είχα άλλε υποχρεώσεις, δεν μπόρεσα να πάω, τα είχα ακυρώσει, τέλο πάντων. Ε, το να αποκλείονται οι δημοσιογράφοι και μετά να λέμε ότι έτσι αποφασίστηκε ο προπολογισμό, είναι αδύνατο να γίνει. Είναι αδιανόητα πράγματα. Δηλαδή εδώ ε, ποδοπατούν Βασικέ αρχέ τη δημοκρατία. Πρέπει να πάρουμε θέση σαφή. Στο παρελθόν πάντοτε το κάναμε. Το πώ θα αποφασίσουμε είναι άλλο θέμα, αλλά δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τα πράγματα βαίνουν ω συνήθω business as usual, για να πάμε να δούμε τα κόμματα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ούτε μπορεί κανεί να μεταχειρίζεται με αυτόν τον τρόπο την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Πρέπει λοιπόν, είμαστε υποχρεωμένοι να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα και να στείλουμε σαφή μηνύματα. Και τώρα η κυρία Γιανακουδάκη. Ευχαριστώ κυρία Κρέμερ. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στα δικαιώματα των ΛΟΑΔ. Νομίζω ότι αναφέρθηκε ότι ήταν αδύναμη αυτή η πτυχή. Κάτι παραπάνω θα έλεγα. Το 2004 ε, υπήρξε θεώρηση της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων και απομακρύνθηκε, καταργήθηκε η αναφορά στο γενετήσιο προσανατολισμό. Ε, ουσιαστικά αναφέρθηκαν ε, σε γάμους που γίνονται μεταξύ ζώων και εγώ το θεωρώ αυτό πολύ αρνητικό σημαντικό επίσης για την Gay Parade του 2013. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι υπάρχει πάρα πολύ λίγη υποστήριξη από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα που έχουν η ΛΟΑΔ. Νομίζω ότι πρέπει να υποστηρίξει αυτό το κοινοβούλιο κάτι τέτοιο και να ζητήσουμε από τις αρχές της ΦΥΡΟΜ ότι η εκδήλωση θα λάβει χώρα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αλαβράκος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ως αντιπρόεδρος της, ε, του υψηλού επίπεδου ε, Επιτροπής για την ΦΥΡΟΜ χαίρομαι ιδιαίτερα να ακούω ότι οι εξελίξεις στα ανθρώπινα δικαιώματα βαίνουν βελτιούμενες. Το θέμα είναι εάν και κατά πόσον η βελτίωση αυτή είναι ικανή να φτάσει στις παρυφές των απόψεων που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα ή εξακολουθούν να μένουν μακριά. Το σίγουρο ξέρετε είναι ότι όταν απογειώνεται ένα αεροπλάνο δείχνει ότι ανεβαίνει πόντους, ανεβαίνει μέτρα, ανεβαίνει ε, σε μια σταθερή πορεία. Φοβάμαι ότι ακόμη είναι στο ανέβασμα η χώρα αυτή και δεν έχει φτάσει σε μια τροχιά ε, ίσης γραμμής. Ε, και το λέω αυτό γιατί η διαφθορά έχει παραμείνει, το, έχει το δικαστικό σύστημα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα, η διαφθορά είναι εντονή, οι κανόνες αγοράς δεν έχουν περάσει και μάλιστα δυστυχώς η διαφθορά ήταν τόσο εντονή ώστε εστέρισαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόπερση ε, από τον εισηγητή για την ε, ενταξιακή πορεία της ΦΥΡΟΜ τον κύριο Τάλερ, ο οποίος πλάκη πιστεύω αθελάτου σε ένα σκάνδαλο για το οποίο κατεδικάστη ήδη προχθές σε τέσσερα χρόνια φυλακή ένας αυστριακός συναδελφός μας. Ε, έχω ζητήσει διαρεύνηση έκτοτε του γεγονότος κατά πόσον υπήρξε θέμα χρηματισμού που συνδέεται με την ΦΥΡΟΜ ή αλλά ακόμη φαίνεται ότι η πορεία της υποθέσεως δεν έχει φτάσει ε, στο σημείο κάποιου πορίσματος. Θα είμαι ιδιαίτερα ευτυχής να μην συνδέεται με τη Φύρο. Εκείνο το οποίο θέλω να πω σε σχέση με το ταξίδι το οποίο προγραμματίζουμε είναι το δίλημα η μετάβασή μας εκεί θα εκλειφθεί ως μποϊκοτάρισμα του Ευρωκοινοβουλίου ή ως φιλοκυβερνητική ενέργεια. Αυτό είναι το στοιχείο το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει ιδιαίτερα και να δούμε εάν πάμε εκεί η κοινή γνώμη, η κυβέρνηση πώς θα χρησιμοποιήσει το θέμα. Θα μας φέρει σε αντίθεση με την αντιπολίτευση, θα το θεωρήσει φιλοκυβερνητική στήριξη. Εάν δεν πάμε εκεί, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Κούκαν, γιατί και εγώ εναντίον των ε, αποκλεισμών των ε, κοινοβουλίων δεν είμαι, μήπως θεωρηθεί ότι κάνουμε κατά κάποιο τρόπο αποκλεισμό του κοινοβουλίου. Πρέπει όμως να λάβουμε ιδιαίτερα υπόψη μας ότι η περιοχή και οι απόψεις στην περιοχή είναι ιδιάζουσες. Αυτά ήθελα να πω και νομίζω ότι αύριο που θα αποφασίσουμε τουλάχιστον εμείς στην Επιτροπή τη μετάβαση θα ανταλλάξουμε τις απόψεις. Θα χαρώ ιδιαίτερα πάντα να πηγαίνει καλύτερα η ΦΥΡΟ. Ευχαριστώ. Okay. Thank you. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να αναφέρω ότι από την ε, πρεσβεία βρίσκεται εδώ η κυρία Γιάσνα Μπολιάτ που έχει προετοιμάσει μια γραπτή δήλωση, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής μας και η ΛΥΠΗ θα λάβουν τη δήλωσή σας σε γραπτή μορφή. Για καταλαβαίνω είναι ιδιαίτερα λεπτομερής. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Άκουσα μόνο μια συγκεκριμένη ερώτηση από τον κύριο Κράμερ στην Επιτροπή. Κύριε Κράμερ, ε, συμφωνείτε διμερώς να σας δοθεί η απάντηση, γιατί πραγματικά μου καθυστερήσει πάρα πολύ. Και για το θέμα των ε, ΛΟΑΔ θα συνεχίσει να εργάζεται η αντιπροσωπεία. Όχι, ας μου πει κανεί μόνο αν υπήρξε αντίδραση, ναι ή όχι. Εν συντομία. Να μας πείτε αν υπήρξε αντίδραση από την Κομισιόν σε σχέση με τη διάκριση κατά των ε, λεσβιών μου φιλοφίλων, διφιλικών κτλ. Συγγνώμη, αλλά δεν είναι σαφής η ερώτηση για μένα. Μήπως δημερός ε, να μπορέσουμε να τη δούμε. Μάλιστα, μπορείτε να ακολουθήσετε μια γραπτή διαδικασία ή να μιλήσετε μεταξύ σας. Λοιπόν, ο κύριος Χατζημαρκάκης θέλει να πει κάτι. Μια παρατήρηση για όσο είπε ο κύριος Σαλαβράκος. Είναι πάρα πολύ λεπτό το θέμα για το αν θα μεταβούμε ή όχι στη χώρα. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τον προκάτοχο, αυτού που εκπροσωπεί τώρα την Ευρωπαϊκή Ένωση στα Σκόπια, γιατί συνομίλησε με την αντιπολίτευση και το... ήταν εν persona non στη χώρα κατόπιν αυτού ενώ υπηρετούσε την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Εγώ ευχαρίστω να δω εσά ω αντιπρόεδρο και τον κύριο Κράμερ για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, γιατί μπορεί να υπάρχουν και άλλε δυνατότητε. Δηλαδή να πάμε όχι υπό την ομπρέλα τη JPC, τη Κοινοβουλευτική Επιτροπή, αλλά μια άλλη ιδιότητα. Θα το συζητήσουμε και θα σα ενημερώσουμε. Μάλιστα, σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και για τη συνεργασία και στην περίπτωση που ταξιδέψουμε φέτος ε, να δούμε με ποιους φορείς θα έχουμε μια κοινή συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο που αφορά την Αιθιοπία. Σας παρακαλώ οι προσκεκλημένοι να έρθουν εδώ στο πάνελ και να δούμε αν μπορούμε να έχουμε και λίγο περισσότερο χρόνο για τη συζήτηση. Uh, um, λοιπόν, συνάδελφοι, να αλλάξουμε λίγο τη σειρά της συζήτηση. Θα δούμε το βίντεο στο τέλος, γιατί δεν χρειαζόμαστε τη διερμηνία για το βίντεο. Ξέρετε ότι αποφασίσαμε... Σας παρακαλώ, όσοι δεν παρακολουθείτε τη συζήτηση για την Αιθιοπία, να αποχωρήσετε. Ευχαριστώ. Θα στείλουμε μία αντιπροσωπεία ντρουά στην Αιθιοπία από τις 10 στις 14 ε, Φεβρουαρίου και καλούμε την αντιπροσωπεία να ε, συναντήσει μια ολοκληρωμένη την Αφρικανική Ένωση και την επόμενη μέρα να επικεντρωθεί στην κατάσταση στην Αιθιοπία. Και όταν λέω εμείς, αυτή τη στιγμή έχουμε τρία άτομα που θα πάνε ο κύριος Ροάτα, ο αντιπρόεδρος της Ντρουά, εγώ, υποφαινόμενη και Δυστυχώ δεν είναι σαφέ ποιο θα είναι το τρίτο άτομο. Ποιο θα είναι το τρίτο άτομο. Ελπίζω να βρούμε κάποιον. Διαφορετικά θα πάμε εμεί οι δύο. Βέβαια έχουμε μεγάλη εμπειρία με διάφορες ε, αποστολές ε, των εκλογών στην Αιθιοπία αλλά οργανώσαμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων γιατί θέλουμε να έχουμε και άμεσες πληροφορίες επικεντρωνόμενοι μόνο στην Αιθιοπία. Για τις άλλες χώρες ε, της Αφρικής θα τα δούμε τα θέματα όταν θα προετοιμαστούμε για την αποστολή. Έχουμε μαζί μας και από τη Human Rights Watch την κυρία Λέσλι Λεύκοφ Α, συγγνώμη, είχε ένα πρόβλημα με το τρένο η κυρία Λεύκοφ, δεν μπορούσε να είναι εδώ, αλλά έχουμε μαζί μας εμπειρογνώμονα ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έναν ακτιβιστή από την Αιθιοπία που είναι μέλος ε, του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και πρόκειται για τον κύριο Τζέρετ, που θα μας ενημερώσει για την κατάσταση τη κοινωνία πολιτών, για την ελευθερία του συνέρχεστα στην Αιθιοπία και για περιπτώσεις ε, ε, υπερασπιστών ανθρωπινών δικαιωμάτων. Και έχουμε και τον κύριο Βίλεμ Όλτχοφ από την ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑΝΤΕΒΚΟ που θα μας ενημερώσει για ε, κάποια project που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση επί τόπου. και από την Υπηρεσία εξωτερική Δράσης είναι εδώ η κυρία Φραντσέσκα Ράτο από το Αιθιοπικό Desk Office. Και βλέπω και τον κύριο Βέρμαν. Τον κύριο Μπέρμαν. καλώ ορίσατε. Ήσασταν ε, επικεφαλής ε, της ε, αποστολής παρατήρησης των εκλογών το 2010 η κυρία Γκόμε είναι τακτικό μέλο, συνεργό, χαίρομαι που είστε εδώ, αλλά δεν θα σα καλωσορίσω ειδικά. You, you what? Oh, Σχόλια εκτός μικροφώνου. Το 2005, μάλιστα, αλλά δεν επικεντρωνόμαστε τόσο στις εκλογές. Θα επικεντρωθούμε στα ανθρώπινα δικαιώματα. Βλέπουμε εδώ και εκπρόσωπο από την Αιθιοπία και σας ευχαριστούμε. Να ξεκινήσουμε με εσά. Uh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πριν να σας δώσω την μαρτυρία μου, θα ήθελα να κάνω μια μικρή παρατήρηση σε αυτήν την παρουσίαση. Δεν εκπροσωπώ το Αιθιοπικό Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αν και ήμουν μέλος του προσωπικού του στο παρελθόν και έχω εργαστεί επί 8 χρόνια. Γι' αυτό σήμερα ζω εξόριστος εδώ, εξαιτίας ίσως της συμμετοχής μου. Επομένως μιλώ με ε, ιδιότητά μου ως μεμονωμένο πρόσωπο. Δεν εκπροσωπώ κανέναν αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία για δεύτερη φορά να απευθυνθώ σε εσά και να εκφράσω τι ανησυχίε μου για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αιθιοπία. Σε αυτήν τη σημαντική ακρόαση έχουν περάσει σχεδόν 7 χρόνια από τότε που είχα δώσει για πρώτη φορά την μαρτυρία μου στην ε, έκτακτη συνάντηση τη Επιτροπής Ανθρωπίνων, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου. Τότε ήταν 15 Μαου 2005. Είχα μιλήσει για τις πολιτικές δολοφονίες περίπου 200 αθώων αμάχων στους δρόμους της Αντιζάπαμπα. Σήμερα θέλω να μιλήσω για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αιθιοπία, κυρίως όσον αφορά την ελευθερία της, του συναθρίζεστε και την ελευθερία του τύπου. Τα 7 χρόνια που μεσολάβησαν από, μετά τις εκλογές του 2005 κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αιθιοπία έχει αλλάξει άρδιν, όχι προς το καλό. Το μοτίβο αυθαίρετης πολιτικής καταπίεσης και παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υπήρχε στην χώρα έχει ε, τώρα μετατραπεί, μεταμορφωθεί μέσω ενός νέου νομικού πλαισίου έχει υιοθετηθεί ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο παρέχει στις κυβερνητικές αρχές αυθαίρετα ε, αυθαίρετες εξουσίες κατά παράβαση των διεθνών προτύπων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα τελευταία έξι χρόνια το Αιθιοπικό Κοινοβούλιο, ιδίω μετά τις εκλογές του 2010, στις οποίες το κυβερνών κόμμα έλαβε ποσοστό 99,6% το κοινοβούλιο λοιπόν αυτό έχει λάβει δρακόντρια ε, μέτρα και νομοθεσία κυρίως για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και για τον περιορισμό της λειτουργίας της κοινωνίας των πολιτών. Η στρατηγική της κυβέρνησης είναι να ελέγχει τον τύπο και οποιονδήποτε πολιτικό αντίπαλο. Η Αιθιοπία είναι μια χώρα στην οποία ε, οι δημοσιογράφοι πέφτουν θύματα των ε, νόμων κατά της τρομοκρατίας και, της, και, και υφίστανται διώξεις από την κυβέρνηση. Το ιστορικό της ε, Αιθιοπίας στον τομέα αυτό είναι εξαιρετικά άσχημο. 79 δημοσιογράφοι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα από το 2001 μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την Διεθνή Επιτροπή Δημοσιογράφων, και αυτό επειδή φοβούνται να πέσουν, μήπως πέσουν θύματα βασανιστήριων, παράνομης κράτησης, ή να υποστούν κακομεταχείριση. Πολλέ φορέ έχουν συμβεί τέτοια περιστατικά με δημοσιογράφου, έχουν, υπο... έχουν επίση υποστεί, δεχθεί και απειλέ κατά τη ζωή του. Οι δημοσιογράφοι αντιμετωπίζουν κατηγορίε για τρομοκρατία και αναγκάζονται να καταλήψουν τη χώρα. Σύμφερα με την εκτίση έκθεση τη ε, ε, Διεθνού Ένωση Δημοσιογράφων του 2012, αγνοούνται δύο δημοσιογράφοι από την Αιθιοπία Του οποίου το 2007 τον Απρίλιο ο Ιθίωπα υπουργό Εξωτερικών είχε παρουσιάσει στην κρατική τηλεόραση ως υπόπτου για τρομοκρατία. Τα, οι τέσσερι αυτοί Αιθίωπες δημοσιογράφοι είναι οι εξή Ρεγιώτα Λεμού, Εσκίντερ Νέγκα, Πουσπέταγε και Ιουσούφ Κετατσιού. Ο κύριο Αλεμού αρθρογραφούσε στην εφημερίδα Φετέχ, που σήμερα έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία της από την αιθιοπική κυβέρνηση, καθώς ήταν επίσης ε, δάσκαλος σε γυμνάσιο, σε λύκειο στην Αντισάπαμπα. Συνελήφθη 21 Ιουνίου του 2011 και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τρομοκρατία το επιθέσεις του Σεπτεμβρίου, το Σεπτέμβριο του 2011. Τον Ιανουάριο του 2012 καταδικάστηκε σε 14 χρόνια ε, φυλάκιση και σε περίπου 1.200 ευρώ πρόστιμο. Τον Αύγουστο του 2012 εκδικάστηκε η υπόθεση στο εφετείο, δεν βρέθη κανένα δικονομικό πρόβλημα και επικυρώθηκε η πενταετής του κάθριξη. Ο Εσκίντερ Νεγκά ήταν μπλόκερ και δημοσιογράφος, είναι μπλόκερ και δημοσιογράφος στην Ιθιοπία, αντιμετωπίζει παρόμοιες κατηγορίες, συνελήφθη το 2005, κατηγορήθηκε για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και για συνωμοσία, του Άλλοι τέσσερι ε, δημοσιογράφοι που βρίσκονταν σε ε, που εξόριστοι κα, ε, καταδικάστηκαν μαζί με τον Νεγκά στη δίκη του. Το δικαστήριο επίσης αποφάσισε την κατάσχεση του σπιτιού του και του αυτοκινήτου της γυναίκας του. Ο Βουσπεταϊέ, δημοσιογράφο δημοσιογράφος στην Αουράμπα Times. Επίσης συνελήφθη 19 Ιουνίου του 2011 με την κατηγορία της ε, προετοιμασία τρομοκρατικού ε, χτυπήματο. Ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας, ο κύριος Κεντέρε, κατάφερε τον ε, Νοέμβριο του 2011 να διαφύγει της χώρας πριν να του απαγγελθούν κατηγορίες με, βάση τον νόμο καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Ο κύριος καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκιση κατά τη διάρκεια της κράτησής του υπέστη βασανιστήρια. Ο κύριος Ιουσούφ Κετατσέ αρθρογραφούσε στην Μουσλιμο Κουτάι συνελήφθη 20 Ιουλίου 2012 και μεταφέρθηκε στο κέντρο κράτησης Μακελάι τον Οκτώβριο του 2012 απαγγέλλονται ε, κατηγορίες με βάση τον νόμο ε, κατά της τρομοκρατίας και σύμφωνα με τις ε, αναφορές της Παγκοσμίας Ένωσης Δημοσιογράφων έχει υποστεί βασανιστήρια στην φυλακή. Και άλλοι δημοσιογράφοι, τοπικοί δημοσιογράφοι, υφίστανται διώξεις και κινδυνεύουν. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση της εβδομαδίας εφημερίδας ΦΕΤΕΧ κατά τις οποίες ασκήθη δίωξη για συκοφαντική δυσφήμιση τον Αύγουστο του 2012. Ο αρχισυντάκτης της κρατήθηκε για ορισμένες μέρες μετά αυτή την άσκηση δίωξης. Τώρα περνώ στο ζήτημα του ε, ελευθερίας του συναθρίζεστε. Ο, ο νόμος 621 του 2009 που υιοθέτησε τον Ιανουάριο του 2009 το Αιθιοπικό Κοινοβούλιο περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα των ε, οργανώσεων ε, των φιλανθρωπικών και των ε, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ιδιαίτερα εκείνων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν θα πω στις λεπτομέρειες των συγκεκριμένων περιορισμών που τίθενται μέσω αυτού του νόμου αλλά το αποτέλεσμα, ο αυτής, αλλά θα μιλήσω για τον αντίκτυπο αυτής της νομοθεσίας μετά την υιοθέτησή της. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασία τον το Νοέμβριο του 2012, η Αιθιοπία είναι μία από τις πέντε χώρες στι οποίες διαπιστώνεται σοβαρή, παραβιάσει τη παραβιάσεις του συναθρίζεσαι. Μετά από την υιοθέτηση αυτή τη νομοθεσία, πολλοί υπερασπιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα. Σημαντικέ οργανώσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων επίση έχουν αναγκαστεί να αυτολογοκρίνονται για να αποφύγουν τις, διμενές, τις αυτή επιπτώσεις αυτής της νομοθεσίας. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας το 2012, τουλάχιστον 17 οργανώσεις άλλαξαν το πεδίο δραστηριότητάς τους και δεν μιλούν πλέον για ανθρώπινα δικαιώματα, μιλούν για αναπτυξιακή συνεργασία. Η σημαντικότερη και μόνη οργάνωση στην Αθιοπία η οποία προσπαθεί να παρακολουθεί τις εξέλιξεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, το Αιθιοπικό Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναγκάστηκε να αλλάξει την επωνυμία του ε, με τη διαδικασία επανακαταγραφής του στα Μητρώα. στην νομοθεσία προβλέπεται ότι δεν έχουν το, το, το, το, δικαίωμα, δεν έχει το δικαίωμα καμιά οργάνωση να χρησιμοποιεί τη λέξη εφιοπία στην επωνυμία της εάν δεν έχει τουλάχιστον πέντε περιφερειακά γραφεία. Επίσης αναγκάστηκε να απολύσει τουλάχιστον έξι μέλη του προσωπικού. Τον Δεκέμβριο του 2009 ε, το, η κυβέρνηση διέταξε να ε, παγώσουν οι λογαριασμοί του Συμβουλίου και περίπου 9,5 μπυρ, ηθιοπικά μπυρ, δηλαδή περίπου 500.000 ευρώ. Μια άλλη σημαντική οργάνωση, η Αιθιοπική Ένωση Γυναικών Δικηγόρων, η οποία δημιουργήθηκε το 1995, επίσης αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα. Αναγκάστηκε να απολύσει το 70% του προσωπικού του το 2010 και το 2011 ενώ ταυτόχρονα τα περιουσιακά στοιχεία της έχουν παγώσει. Έχουν δεσμευτεί. Το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε την έφεση που άσκησε αυτή, η Ένωση. Επομένως παραμένουν δεσμευμένα τα περιουσιακά στοιχεία της. Και τέλος, η, η, η Ένωση Αιθιώπων ε, διδασκάλων ένα σημαντικό συνδικαλιστικό σωματείο δεν έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί στα Μητρώα με βάση τη νέα νομοθεσία. Λοιπόν, συμπερασματικά, η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει επιδεινωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια. Η κυβέρνηση επιδιώκει να περάσει ένα, να δημιουργήσει ένα νομικό, και θεσμικό πλαίσιο το οποίο να δικαιολογεί και το οποίο να τη δίνει τη δυνατότητα να συνεχίζει τι παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αντί να τι αντιμετωπίσει, αντί να ε, ξεκινήσει μια προσπάθεια εκδημοκρατισμού και εμπέδωση του κράτου δικαίου. Ω αποτέλεσμα, χιλιάδε Αιθίωπε εγκαταλείπουν τη χώρα κάθε χρόνο. Άλλοι κρατούνται ε, επιμακρών εξαιτία των πολιτικών του πεπιθήσεων ή των απόψεων που εξέφρασαν. Οι οργανώσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι υπερασπιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οργανώσει τη κοινωνία των πολιτών δεν απολαμβάνουν ελευθερία τη έκφραση, δεν απολαμβάνουν ελευθερία του συναθρίζεσθε. Ταυτόχρονα δεν, δεν υφίσταται στην Αιθιοπία καν το δικαίωμα τη ειρηνική διαδήλωση. Είναι καλό παράδειγμα πιστεύω η βίαιη καταστολή του κινήματος των Αιθιώπων μουσουλμάνων, των ειρηνικών διαδηλώσεών τους από την κυβέρνηση. Οι κυβερνητικοί ε, αξιωματούχοι ε, και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας συνέλαβαν και υπέβαλαν σε κακομεταχείριση τα, ε, αυτούς τους ειρηνικούς διαδηλωτές. Παραμένουν πολλοί από αυτούς κρατούμενοι και τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες με βάση τον νόμο περί τρομοκρατίας. Ο νόμος περί τρομοκρατίας δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να κρατά ανθρώπους χωρίς να έχουν ασκήσει καμία πράξη βίας. Τις περισσότερες φορές το μόνο τους έγκλημα είναι ότι εξέφρασαν τις πολιτικές τους πεπιθήσεις ή άλλες πεπιθήσεις τους και ότι άσκησαν κριτική στην πολιτική και τις πρακτικές της κυβέρνησης. Ευελπιστώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η αποστολή της Επιτροπής σας θα προσπαθήσει να διαπιστώσει την κατάσταση επιτόπου, την κατάσταση όπως σας την περιέγραψα και συμπερασματικά θα ήθελα να προτείνω έντονα στην αντιπροσωπεία σας να συναντηθεί, να επιδιώξει να συναντηθεί με αυτούς τους τέσσερις φυλακισμένους δημοσιογράφους στην Αιθιοπία και να συνομιλήσει με οργανώσεις και υπερασπιστές των ανθρωπινών δικαιωμάτων που έχουν, δεν έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Χαλέ Μαριά μου για τη δήλωση αυτή και τις ε, συστάσεις προς εμάς. Και τώρα ο κύριος ε, Ολτσχόφα από την Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ θα μας ε, μιλήσει και για κάποια ε, χρηματοδοτούμενα από την Ένωση προγράμματα. Μπορούμε να επισκεφθούμε. Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε, μου ζητήθηκε συγκεκριμένα να μιλήσω για τη συνεργασία με τις οργανώσεις ε, της κοινωνίας των πολιτών και γι' αυτό καλό θα ήταν να δώσω κάποιο ιστορικό υπόβαθρο για τον νόμο για τις οργανώσεις αυτές που αναφέρθηκε. Ο νόμος ε, αφορά φιλανθρωπικές οργανώσεις ε, και εταιρείε. Είναι από το 2009 νόμος που προβλέπει τα δικαιώματα φιλανθρωπικών οργανώσεων και υποχρεώσεις τους. Ο νόμος αυτός προβλέπει μια καινούργια υπηρεσία για τις ε, φιλανθρωπικές ε, οργανώσεις και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και όλες πρέπει να καταχωρίζονται εκεί, στην υπηρεσία. Μεταξύ άλλων παρακολουθεί η υπηρεσία των τομέα και υποβάλλει εκθέσεις στην κυβέρνηση. Αυτή η υπηρεσία επίσης δίνει κατευθυντηρίες γραμμές, οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου. Αυτό που είναι σημαντικό στο νόμο είναι ότι υπάρχει και μια κατηγοριοποίηση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε τρεις κατηγορίες. Υπάρχουν ξένες φιλανθρωπικές οργανώσεις, μετά έθιοπικές, με στην Αιθιοπία, οργανώσεις που λειτουργούν με πάνω από το 10% των εισοδήματων από ξένες, των εσόδων τους από ξένες πηγές και τρίτον αιθιοπικές ε, οργανώσεις. Αυτές της τρίτης κατηγορίας δεν μπορούν να παίρνουν πάνω από το 10% των εσόδων τους από ξένες πηγές. Τώρα δράσεις για την ευαισθηκοτοποίηση και αλλού γίνεται επιτρέπεται μόνο για την τρίτη κατηγορία, τις αιθιοπικές. Επίσης, είναι σημαντικό για να κατανοηθεί το θέμα να αναφέρουμε μια κατευθυντήρια γραμμή από τον Ιούλιο του 2011, η οποία καθορίζει διοικητικό και λειτουργικές δαπάνες των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Είναι η κατευθυντήρια γραμμή ως 3070 λέει ότι το διοικητικό κόστος δαπάνες μιας εταιρείας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30% των συνολικών δαπανών και η ιδέα είναι ότι τα περισσότερα κονδύλια πρέπει να πηγαίνουν στην εφαρμογή. Ε, έχει ευρία κάλυψη το διοικητικό κόστος και γι' αυτό είναι δύσκολο να εφαρμοστεί από τις οργανώσεις, πολλές από τις οργανώσεις και τα δίκτυα των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών αυτή η κατευθυντήρια γραμμή. Παρουσίασα αυτό το νομικό πλαίσιο εν ολίγης για να δώσω ο, κάποιες πληροφορίες για το πώς συνεργαζόμεθα στην Αιθιοπία με αυτές τις οργανώσεις, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για κονδυλία από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Εδώ και κάποια χρόνια υπάρχει εν λειτουργία το λεγόμενο Ταμείο για την Κοινωνία των Πολιτών. Το πρώτο ταμείο ε, καλύφθηκε από το ένατο ταμείο και είχε 8,5 εκατομμύρια. Λειτουργούσε μέχρι το 2011 και οι εμπειρίες ήταν πολύ θετικές, η αξιολόγηση ήταν θετική, πολύ σημαντικό, πολύ αποδοτικό, πολύ αποτελεσματικό. Αλλά αυτά ήταν πριν από την θέση σε ισχύ της νομοθεσίας για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Με τον καινούριο νόμο υπάρχει συνέχιση της υποστήριξης των οργανώσεων αυτών στα πλαίσια του 10ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης και δώσαμε σε διαβούλευση με την Αιθιοπική Κυβέρνηση περισσότερα κονδύλια στο Ταμείο. Υπάρχουν δύο φάσεις. Ε, κάθε μία από 6 ε, εκατομμύρια, 12 συνολικά. Η πρώτη φάση άρχισε πέρσι, το 2012. Η δεύτερη φάση προγραμματίζεται για το 2013 και αυτό θα έχει αποτέλεσμα το 2014. Αυτό το Ταμείο για την Κοινωνία των Πολιτών είναι λίγο μοναδικό. Η χρηματοδότηση αναφέρεται ως εγχώρια, η εθνική, η εσωτερική. Όλες οι οργανώσεις αυτές της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να υποστηριχθούν από αυτά τα ταμεία όπως και οι οργανώσεις που αφορούν θέματα διακυβέρνησης, δηλαδή οι έθιοπικές οργανώσεις και υπηρεσίες και φιλανθρωπικές οργανώσεις. Το πρόγραμμα έχει δύο συνιστώσεις. Από τη μία πλευρά ε, δίνονται χορηγήσεις στις οργανώσεις αυτές ε, μέσα από προσκλήσεις υποβολή προτάσεων σε διάφορους τομείς συνεργασίας με την Ένωση και την Αιθιοπία περιλαμβάνοντας ε, δημοκρατική διακυβέρνηση, πρόσβαση στη δικαιοσύνη, περιβάλλον και άλλα. Και από την άλλη υπάρχει τεχνική υποστήριξη, όχι επιχορηγήσεις, για την εκπαίδευση, και παρακολούθηση των μη των οργανώσεων αυτών σε θέματα ηγεσία, λογοδοσία, ε, ένταξη ε, τη διάσταση του κοινωνικού του φύλου. Υπάρχει και μια τριμερής ε, διευθύνουσα επιτροπή για τα προγράμματα που αποτελείται από εκπροσώπους της κυβέρνησης, της κοινωνίας των πολιτών και της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η πλειοψηφία των εδρών σε αυτή την Διευθύνουσα Επιτροπή είναι από τα μέλη της Επιτροπής των Οργανώσεων αυτών ε, για να προωθηθεί ο διάλογος και η εμπιστοσύνη μεταξύ των τριών μερών, γι' αυτό τριμερής. Υπάρχει ένα πρόγραμμα στο οποίο δραστηριοποιούμεθα για να στηρίξουμε την κοινωνία των πολιτών στην Αιθιοπία με στόχο να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε μια σφίζουσα κοινωνία των πολιτών στη χώρα αυτή δυναμική που θα συμμετέχει και στη συμμετοχική δημοκρατία σε όλες τις εκφάνσεις και στην ανάπτυξη. Ένα δεύτερο πρόγραμμα όπου η ενωσιακή συμμετοχή είναι αξιόλογη είναι ένα πρόγραμμα προώθησης των βασικών υπηρεσιών. Μεγάλο πρόγραμμα με πολλούς δωρητές που υποστηρίζεται και από την Παγκόσμια Τράπεζα και από την Αφρικανική Τράπεζα, ε, την Αυστρία, την Ιταλία, την Αφρικανική Τράπεζα ανάπτυξη, Είναι ένα πρόγραμμα για να ε, μεταδώσει βασικές υπηρεσίες στην εκπαίδευση, την υγεία, την ε, ίδρευση, ε, την ε, υποδομή σε όλη τη χώρα, υποδομές. Και Υπάρχει και ένα στοιχείο κοινωνική ευθύνη και λογοδοσία που εφαρμόζεται από τι οργανώσει τη κοινωνία των πολιτών, CSOs όπω λέμε, οι οποίε συμμετέχουν σε εκστρατείε ε, ευαισθητοποίησης για τις διάφορες δραστηριότητες, σχεδιασμός, ε, ε, κατάρτιση προπολογισμού, σε τοπικό επίπεδο και θέματα που αφορούν την λογοδοσία και τι καταγγελίε. Τα ταμεία που στηρίζουν τις CSOs θεωρούνται εθνική χρηματοδότηση και αυτά και διάφορες CSOs μπορεί να ε, υποστηριχθούν από εκεί. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα θέματα υποστήριξης των CSOs, ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ της κυβέρνησης και των τομέων CSOs. Αυτά όμως θα τα πούν οι ε, συνάδελφοι από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ και για τη λεπτομερή περιγραφή. Νομίζω ότι όλοι όσοι ενδιαφερόμαστε μπορούμε να έχουμε αυτά τα στοιχεία και γραπτός. Παρακαλώ από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Έχετε το λόγο. Ναι, καλησπέρα σε όλους ε, και σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε σε αυτή τη συνεδρίαση. Μου δίνετε τη δυνατότητα να συμπληρώσω αυτό που είπε ο συνάδελφος από την ΤΕΦΚΟ. Θα επιβεβαιώσω καταρχήν ότι πράγματι ανησυχεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία της συνοχής και το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως η αντιτρομοκρατική νομοθεσία η Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά αναγνωρίζει τα, τις προκλήσεις της τρομοκρατίας που αντιμετωπίζει η Αιθιοπία και νομιμείται η κυβέρνηση να την καταπολεμήσει όμως μπορεί να έχει ε, αντίκτυπο η νομοθεσία αυτή στην ελευθερία της έκφρασης αν ερμηνευτεί ευραίως. Έτσι λοιπόν η προσθέμενη εξέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταρχήν είναι όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά να υπάρξει και συμπληρωματική δράση με τα κράτη-μέλη. Έχουμε 20 κράτη-μέλη στην Αιθιοπία. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους αριθμούς εκπροσώπησης στην Αφρική και ουσιαστικά επιβεβαιώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι υπάρχουν πολλαπλή τρόποι διαλόγου και συνεργασίας. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται σε καλά προσδιορισμένες πολιτικές για το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, θέτοντας ένα πλαίσιο για την υλοποίηση των εργασιών. Επίσης, η στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση Αφρική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να πλαισιώσει τις διμερείς σχέσει σε ένα πιο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Πιο συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Ένωση ω ε, ομάδα συγκέντρωσης μέσων, ε, όπως ε, είπατε κι εσείς, η ανθρωπιστική παρέμβαση μπορεί να συνδυαστεί με διπλωματικές δράσεις. Έτσι λοιπόν Είμαι στη διάθεσή σας ε, για οποιασδήποτε περαιτέρω ερωτήσεις έχετε. Πέντε κυρίες δράσεις νομίζω ήταν πάρα πολύ σημαντικές. Καταρχήν, ο τομέας της κοινωνίας των πολιτών, η σχετική ομάδα εργασίας, ε, η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε αυτή την ομάδα εργασίας το 2012. Εκεί συμμετέχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης και της κοινωνίας των πολιτών και των δωρητών συμπροεδρεύει ο Υπουργό Εκτορικών Υποθέσεων ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και της τη Εθνοπίας ήδη συναντήθηκε πέντε φορές το 2012 και σύμφωνα στην αντικοποίηση τη εργασία τη το 2013 με μηνιαίε συνεδριάσεις. Πρόκειται για ένα φόρουμ όπου ο αντίκτυπος ε, της ε, κοινωνίας ε, των πολιτών και οι κατευθυντήριε γραμμέ για την κοινωνία των πολιτών συζητούνται. Επίση έχουμε το φόρουμ υψηλού επίπεδου μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών και Οικονομικής Ανάπτυξης ε, και έχουμε εκεί τη συμμετοχή, μάλλον έχουμε ε, το θέμα της κοινωνίας των πολιτών, υπάρχει στην για διάταξη από το 2010 και ε, εκεί έχουν προσθεθεί και νέα θέματα στην ευρωπαϊκή διάταξη. Τρίτην, έχουμε το Ταμείο Ευρω... ε, της Κοινωνίας των Πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση που στήθηκε το 2010 και ο συνολικό στόχο ήταν να αυξηθεί και να βελτιωθεί ο ρόλος των μη κρατικών φορέων έτσι ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή και συνεισφορά των οργανώσεων τη κοινωνία των πολιτών σε βασικού τομεί διακυβέρνηση και ανάπτυξη. Επιπλέον, έχουμε άλλο ένα φόρουμ ανταλλαγή απόψεων μεταξύ κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, έχουμε ε, το σχετικό άρθρο της, ε, που βασίζεται στο σχετικό άρθρο της Συμφωνίας του Κοτονού. Η πιο πρόσφατη συνάντηση που είχαμε, δυνάμει του διαλόγου του άρθρου Α, ήταν με τον νέο Πρωθυπουργό, λέμε από το προηγούμενο Δεκέμβρη, 13 Δεκεμβρίου 2012. Κατά την ε, τελευταία συνεδρίαση πολιτικού διαλόγου μεταξύ άλλων θεμάτων, η Ευρωπαϊκή Ένωση συζήτησε και θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τον Πρωθυπουργό. Ήταν μια ανοιχτή συζήτηση και θέσαμε συγκεκριμένα δύο ζητήματα. Το ένα αφορούσε ε, την εφαρμογή ε, του ATP, δηλαδή της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας, και το άλλο θέμα αφορούσε τους παγωμένους λογαριασμούς δύο ακτιβιστών ανθρωπίνων, μάλλον δύο ιδρυμάτων, όπου συμμετέχουν ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Αιθιοπία επίσης ε, υποστηρίζονται από την επίτευξη των στόχων της χιλιετίας. Είναι ε, δεσμευμένη να πετύχει τους στόχους αυτούς η κυβέρνηση υποστηρίζοντας και την περιοδική ε, την αναθεώρηση των περιοδικών συστάσεων μπορεί να υπάρχει και ευκαιρία για περαιτέρω εφαρμογή των συνταγματικών αρχών της Αιθιοπίας και ελπίζουμε ότι μαζί με την Αιθιοπία θα υπάρξει δυνατότητα να πάμε περαιτέρω, να πάμε μακρύτερα. Και κάτι τελευταίο και θα σταματήσω εδώ. Νομίζω ότι η αποστολή της Ντρουά στην Αιθιοπία το Φεβρουάριο θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη για να αξιολογήσει την κατάσταση των ανθρωπινών δικαιωμάτων στη χώρα και το πιο σημαντικό για να δείξει ότι υπάρχει παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη δέσμευσή της επιτόπου να στείλει μηνύματα υποστήριξης της πρόθεσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να λάβουμε γραπτό και τη δική σας δήλωση γιατί είχε πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Τώρα, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Μπέρμαν καταρχήν και κατόπιν στην κυρία Γκόμες. Παρακαλώ, κύριε Μπέρμαν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον νούμερο που κατανόμασε αυτούς τους δημοσιογράφους που βρίσκονται στη φυλακή. Είναι πραγματικά τρομερό και για τους δημοσιογράφους αλλά και οποιοδήποτε που έχει καταδικαστεί για πολιτικούς λόγους ε, επειδή έχει εκφράσει την άποψή του σε κάποια άρθρα είναι τρομερό να έχει φυλακιστεί κανείς για το λόγο αυτό και πάντοτε είναι καλό να γνωρίζει κάποιος ότι το όνομά του έχει αναφερθεί δημοσίως κάπου στην Αιθιοπία υπάρχει μια τρομερή καταστολή επί της αντιπολίτευσης, επί των δημοσιογράφων, επί των ακτιβιστών ανθρωπινών δικαιωμάτων και επίσης ε, είναι τρομακτικό ότι οι Ηνωμένες και η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και αν εκτιμώ τις προσπάθειες των συναδέλφων από την Κομισιόν και την, Ευρωπα... την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, οι προσπάθειες να βελτιωθεί η κατάσταση μερικώς είναι τρομακτικό ότι αυτές οι μεγάλες δυνάμεις εξακολουθούν να υποστηρίζουν το καθεστώς. Γιατί το κάνουν αυτό τώρα, λόγω της ε, στρατηγικής θέσεως της Αιθιοπίας στο κέντρο της Αφρικής. Προφανώς ναι. Έχουμε ντρόν ε, που ε, από αμερικανική βάση πετούν στη Σομαλία από την Αιθιοπία. Και Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ κοινικά όλα αυτά και πραγματικά γεμάτα υποκρισία και είναι πραγματικά εκπληκτικό ότι μπορούν να πετάξουν καν αυτά τα ντρόν. Γιατί αν η υποκρισία είχε βάρος δεν θα μπορούσαν να πετάξουν. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι πιο σκληρή στο να καταδικάσει την απόλυτη έλλειψη δημοσίου χώρου και ελευθεριών στη χώρα και θα πρέπει να ζητήσει την απελευθέρωση των πολιτικών ε, κρατουμένων, των δημοσιογράφων που είναι στη φυλακή, να επιμείνει στον υπάρξει ανοιχτό διάλογο με την αντιπολίτευση που δεν έχει καμία δυνατότητα να εκφραστεί με έναν δίκαιο τρόπο. Θα πρέπει να επιμείνει στη μεταρρύθμιση του νόμου περί των πολιτών για τα φιλανθρωπικά ιδρύματα. Θα πρέπει να επιμείνει να θεθεί τέλος στα βασανιστήρια και θα πρέπει να επιμείνει για ε, να ε, γίνουν ε, σεβαστοί κάποιοι άνθρωποι που εξακολουθούν να ζουν σε κάποια χωριά και δεν θέλουν να ζουν σε αστικές περιοχές. Γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ζουν σε πάρα πολύ δύσκολε συνθήκε, σε ημιάγονε περιοχέ. Θα πρέπει να υποστηριχθούν αντί να του στερούν τη γη του. Μιλάμε για 250.000 άτομα περίπου στην Καμπέλα και του αξίζει κάτι καλύτερο. Ε, το 2010 όταν συμμετείχα στην ε, αποστολή παρατηρήσεων των εκλογών δεν έκανα αυτή τη σκληρή κριτική γιατί τότε έπρεπε να ήμουν ουδέτερος και νομίζω ότι η έκθεση που υποβάλαμε ήταν αμερόληπτη, υψηλής ποιότητας και ουδέτερη και θέλω να προστατεύσω την έκθεση αυτή για, δεν θέλω να εκφραστώ με ένα σκληρό τρόπο για το τι συμβαίνει στην Αιθιοπία και πάλι θα συμμετέχω σε διάλογο με τους ηγέτες της Αιθιοπίας. Ε, είμαι ανοιχτό σε κάθε διάλογο, όπως ε, συνομίλησα με τον κ. Ζενάου για ώρε και ώρε και ήταν πάρα πολύ δύσκολη η διαδικασία αυτή. Ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα το αναλάβει αυτό σοβαρά και θα θέσει περισσότερους όρους για την παροχή βοήθειας.